So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Anhörung der designierten Kommission. Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Καλώς ήλθατε στην ακρόαση της υποψήφιας Επιτρόπου για την κλιματική αλλαγή. Θα, θέλω να καλωσορίσω την Κόνη Χέντεγκαρτ στην Επιτροπή μας. Νομίζω ότι γνωρίζετε τη διαδικασία. Καταρχήν θέλω να χαιρετήσω τους εκπροσώπους της Επιτροπής Βιομηχανίας, ο πρόεδρος Herbert Ρόιλιν και αυτός παρόν, επίσης τους συναδέλφους από την Επιτροπή Μεταφορών. Πρόκειται για μια ακρόαση στην οποία εμπλέκονται τρεις διαφορετικές επιτροπές και στις επόμενες τρεις ώρες <clears throat> θα πρέπει το Κοινοβούλιο να σχηματίσει μια εντύπωση σε σχέση με την ε, την δυνατότητα της κυρίας Κόνι Χέντεγκατ να αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της κλιματικής αλλαγής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κρίνει φυσικά και τις ειδικέ γνώσεις της υποψηφίας για το προβλεπόμενο χαρτοφυλάκιο, καθώς και την επικοινωνιακή της ικανότητα, κάτι το οποίο στην ευρωπαϊκή πολιτική είναι πια μεγάλης σημασίας. Αυτές είναι οι κατευθυντήριες γραμμές, αγαπητοί συνάδελφοι, που έχουμε καθορίσει εμείς ήδη για την έγκριση των υποψηφίων επιτρόπων. Στις επόμενες τρεις ώρες θα πρέπει να ακολουθήσουμε τους κανόνες που ήδη σας είναι γνωστοί. Είναι <clears throat> μια διέρεση του χρόνου που πρέπει να παραμείνουμε πιστοί σε αυτήν. Θα δώσουμε το, το λόγο στην κυρία Χέντεγκατ για 10 λεπτά και μετά ακολουθεί η ΚΑΤ επιτραπέζια αντισφαίριση, ανταλλαγή ερωτήσεων και απαντήσεων Έχουμε ένα λεπτό ε, ερώτηση, δύο λεπτά απάντηση, 45 δευτερόλεπτα νέα ερώτηση, ένα λεπτό απάντηση. Όποιο είναι από φυσικά το ερώτημα του εκπίπτει και θέλω να σας τονίσω επίσης ότι η δεύτερη ερώτηση, η συμπληρωματική ερώτηση, θα πρέπει να αναφέρεται στην προηγούμενη ερώτηση. Δηλαδή, δεν είναι ευκαιρία για να θέσει κανεί ένα δεύτερο ερώτημα και έχω φυσικά επιφυλάσσω με το δικαιώματο να απορρίψω μια δεύτερη ερώτηση, αν δεν εμπίπτει σε αυτού του κανόνε. Κυρία Χέντεγκαρτ, Ελπίζω ότι έχετε συνέλθει από τις μαραθώνιες συνεδριάσεις της Κοπενχάγης και εγώ πέρασα μία βδομάδα στις, ε, στην Κοπενχάγη. Ήταν μία αρκετά στρεσαριστική εμπειρία. Έχετε κρατήσει διάφορα αξιώματα. Υπήρξατε υπουργό ε, Περιβάλλοντος και επίσης Υπουργό Κλίματος και Ενέργειας στη χώρα σας και τώρα είστε υποψήφια επίτροπος για την κλιματική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 27 κρατημέρια και 500 εκατομμύρια πολιτών. Γνωρίζετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα τελευταία χρόνια είχε ακολουθήσει ένα, είχε παίξει μάλλον ένα ρόλο κινητήριο σε ό,τι αφορά την κλιματική συζήτηση. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος σας τη της δικής μας Επιτροπής και νομίζω ότι θα το κατανοήσετε και από τις ερωτήσεις που θα σας απευθυνθούν στις επόμενες τρεις ερωτήσεις. Ελπίζουμε λοιπόν ότι <clears throat> θα ακούσουμε από σας κατά τη διάρκεια τη ακρόαση αυτή πώ θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τη μεγάλη απογοήτευση της Κοπενχάγης και να περάσουμε σε νέες ελπίδες για τη διάσκεψη του Μεξικού και επίσης πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δράσει γιατί ξέρουμε ότι αυτά τα οποία έχουμε επιτύχει δεν επαρκούν και επομένως είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πώς θέλετε εσείς να προχωρήσετε για να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς και πώς θα συνεργαστείτε με τους ε, υπόλοιπου επιτρόπους οι οποίοι έχουν σχετικά χαρτοφυλάκια. Αυτά λοιπόν μορφή <clears throat> χαιρετισμού. Κυρία Χέντεγκαρτ και σα δίνω ασμένο τον λόγο. Για 10 λεπτά μάξιμου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι αξιότιμα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, γιατί βρισκόμαστε στην πολιτική. Εγώ νομίζω διότι πιστεύουμε ότι είναι δυνατόν να αλλάξουμε τα πράγματα. Παρά τις διαφορετικές απόψεις και ιδέες, έχουμε όλοι μια κοινή επιθυμία να είναι καλύτερο το αύριο από ότι είναι σήμερα. Νομίζω ότι τα επόμενα πέντε χρόνια πρέπει πολλά να αλλάξουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλιώς, πολιτικά, οικονομικά και στρατηγικά θα υπολοιπόμεθα του υπόλοιπου κόσμου στον 21ο αιώνα. Η πρώτη μου ενσυνείδητη πολιτική δράση ήταν το 1972, όταν ανάρτησα ένα πόστερ στην τάξη μου. Ψηφίστε ναι για την Ευρωπαϊκή κοινότητα. Ο δάσκαλος το κατέβασε κάτω αμέσως. Το 96 ως νέα βουλευτής είπα υποστήριξα το ναι για την ενιαία ευρωπαϊκή πράξη. Βεβαίως και πρέπει να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή συνεργασία. Αργότερα για τα δημοψηφίσματα για το Μάστρι ως δημοσιογράφος ενημέρωσα για τον σκεπτικισμό που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και με χαρά είδα την ιστορική διεύρυνση 10 χρόνια αργότερα που απέδειξε την ανάγκη για μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση και τα τελευταία χρόνια ως υπουργό Περιβάλλοντος και μετά Κλίματος και Ενέργειας είδα από πρώτο χέρι το πόσα μπορούμε να κάνουμε μαζί. Συχνά μάλιστα μπόρεσα να χρησιμοποιήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν μοχλό για εσωτερική δράση. Είχα την τιμή επίσης να συνεργαστώ και με τους ευρωβουλευτές για το REACH, για, την... για τον παροπλισμό πλοίων και άκουσα και τις απόψεις πριν από την COP στην Πότζραν. Ξέρω λοιπόν ποια είναι η αξία να συνεργαζόμαστε στενά και στα έγκαιρα στάδια για να αλλάξουμε τα πράγματα. Και με την προϋπόθεση ότι θα μου δώσετε την ευκαιρία να γίνω η πρώτη επίτροπο για την κλιματική δράση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα χρειαστώ πάντα τις ιδέες σας και την ενίσχυσή σας για να έχουμε υψηλέ φιλοδοξίες. Πώς λοιπόν θα ήθελα να αλλάξει η Ευρώπη μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Θα ήθελα να δω μια Ευρώπη που θα είναι η πιο φιλική προς το περιβάλλον περιοχή του κόσμου και είναι απόδειξη ότι επενδύοντας σε φιλικές και ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες δεν χάνεται αλλά κερδίζεται. Πριν πέντε χρόνια σας είχα πει ότι το 2009 παρά μια ιστορική οικονομική κρίση, κλιματικές αλλαγές θα ήταν στο προσκήνιο της παγκόσμιας ατζέντα τόσο πολύ μάλιστα ώστε 120 αρχηγοί και κρατών και κυβερνήσεων να βρεθούν σε μια διάσκεψη στην Κοπεχάγη, κανένας δεν θα με πίστευε. Και αν σας είχα πει ότι όλοι, όλες οι χώρες που εκπέμπουν θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι για να αναλάβουν κοινή ευθύνη και να επιτύχουν τον στόχο των δύο βαθμών Κελσίου, θα μου λέγατε ότι ονειρευόμουν. Βεβαίως και εγώ απογοητεύτηκα ότι το COP15 δεν έδωσε δεσμευτικούς στόχους. Βεβαίως, πολλά πρέπει ακόμα να γίνουν. Όμως, πολλά άλλαξαν τα τελευταία χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο για να ανοίξει το δρόμο της αλλαγής και μάλιστα ιδιαίτερα για την κοινή γνώμη και την συνειδητοποίηση των θεμάτων αυτών. Τα επόμενα πέντε χρόνια επίσης μπορούν να είναι σημαντική αλλαγή, όχι μόνο εξαιτία των κλιματικών αλλαγών, αλλά και γιατί αν διστάσουμε, αν καθυστερήσουμε, η Ευρώπη θα χάσει την ανάπτυξη, θέσεις απασχόλησης, ευημερίας Είτε υπάρξει διεθνή συμφωνία είτε όχι, η Κίνα προχωρά πολύ γρήγορα. Οι τώρα κατάλαβαν τον μήνυμα και προχωρά πολύ γρήγορα για αποδοτική ενέργεια και τεχνολογία όπως και η Ιαπωνία, η Βραζιλία, η Νότιος Κορέα. Δηλαδή αμφισβητούνται πλέον τα ισχυρά σημεία της Ευρώπης. Πρέπει λοιπόν να ανασυνταχθούμε, να συνεργαστούμε και αν δεν το κάνουμε αυτό χάνουμε. Εάν το κάνουμε έχουμε μια ευκαιρία να κερδίσουμε. Για να εξοικονομήσουμε, το να εξοικονομίζουμε πόρους, ξοδεύουμε, ε, εξοικονομούμε χρήματα. Όταν τα παιδιά μου θα είναι στην ηλικία μου, ο πληθυσμός της γης θα είναι 9 δισεκατομμύρια και οι πόροι θα είναι σπάνιοι. Καθώς επενδύουμε λοιπόν σε βιώσιμο μέλλον, ας επενδύσουμε σε λύσεις που θα είναι προς όφελος του κλίματος, της ενεργειακής ασφάλειας και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν η Ευρώπη είναι πιο έξυπνη στην παραγωγή της και έχει πιο ενεργειακά αποδοτικά ραδιόφωνα από άλλους, όχι μόνο θα είναι προς όφελος του περιβάλλοντος, θα έχουμε λιγότερη ανάγκη να εισαγάγουμε καύσιμα και θα είναι πιθανότατα να έχουμε περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Μπορεί να πούν ορισμένοι ότι δεν, μας, δεν δεν μπορούμε να το κάνουμε. Εγώ λέω ότι είναι απαραίτητο να το κάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ενσωματώσουμε το κλίμα σε όλες τις σχετικές πολιτικές. Για να το επιτύχουμε αυτό θα συνεργαστώ με τους συναδόλφους της Κομισιόν για Μεταφορές, Γεωργία, Βιομηχανία, Ανάπτυξη και βεβαίως και με την ε, Επίτροπο Περιβάλλοντος. Ο κύριος Δήμας είχε μία και μόνη ισχυρή φωνή. Ο κύριος Ποτότσνικ και εγώ θα είμαστε δύο φωνές στο κολέγιο. Όμως όλο, όλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογηθεί για το αν επιτύχει τις πολιτικές κατευθύνσεις γραμμές του Προέδρου Μπαρόζο για τα επόμενα πέντε χρόνια. Η στρατηγική της Λισαβόνας θα πρέπει να προωθέσει τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα, να έχουμε πόρους για αυτές τις έρευνες σε αυτούς τους τομείς και να υπάρξει πολιτική υποστήριξη για την ανάπτυξη νέων πράσινων τεχνολογιών. Είναι αυτονόητο ότι θα εφαρμόσω το συμφωνημένο ενεργειακό και περιβαλλοντικό πακέτο όμως η ενσωμάτωση της πολιτικής αυτής είναι κάτι παραπάνω. Όταν παραδείγματο χάρη μεταρρυθμίζουμε την γεωργία συστηματικά θα πρέπει να ενσωματώσουμε κλιματικές προοπτικές στις προοπτικές μας. Άλλος ένας τομέας είναι οι μεταφορές. Οι εκπομπές που σχετίζονται με τις μεταφορές συνεχώς αυξάνονται και συχνά εξισορροπούν τα όσα επιτυχάνουμε ως μειώσεις σε άλλους τομείς. Υπάρχει νομοθεσία για την μείωση εκπομπών στα αυτοκίνητα, υπάρχει μια πρόταση για να ληφθούν υπόψη οι εκπομπές των αεροσκαφών, αλλά πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα και θα συνεργαστώ με τους ε, επιτρόπους για τις μεταφορές για να έχουμε ένα συνολικό πακέτο. Σε ό,τι αφορά επίσης την προσαρμογή με την μελλοντική συζήτηση για τις δημοσιονομικές προπτικές πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει έλεγχο σε ό,τι αφορά τις κλιματικές επιπτώσεις όλων των προγραμμάτων και υποδομών που εγκρίνονται από την Ένωση. Μόνο έτσι θα έχουμε ολοκληρωμένες στρατηγικές προσαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη σε διεθνές επίπεδο θα, εργαστώ πολύ σκληρά για να έχουμε μια διεθνή αγορά εμπορίας εκπομπών σε όλο τον κόσμο και μέσα στις χώρες του ΟΣΑ μέχρι το 2015 και έχω σκοπό να συσχετίσω το ευρωπαϊκό σύστημα με το αμερικανικό σύστημα ή δυνατόν μέχρι το 2015. Ο προκάτοχός μου εδραίωσε την ευρωπαϊκή αγορά εκπομπών. Μπορεί Τώρα πρέπει να γίνει πιο διεθνές το ευρωπαϊκό σύστημα. Και τέλος υπάρχουν πολλά διδάγματα που μπορούμε να εξάγουμε από την COP15 και είμαι σίγουροι ότι θα έχω την ευκαιρία να επανέλθω σε αυτό το θέμα. Όμως υπάρχουν σημαντικά διδάγματα που πρέπει να εξάγουμε για την Ευρώπη. Τις τελευταίες ώρες στην Κοπεχάγη η Κίνα, η Ινδία, η Ρωσία, η ΙΠΑ και η Ιαπωνία η κάθε μία είχαν μία φωνή ενώ η Ευρώπη είχε πολλές και διαφορετικές φωνές. Μερικές φορές ξοδεύουμε τόσο χρόνο να συμφωνήσουμε μεταξύ μας που όταν τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση φτάσει στις διαπραγματεύσεις της διεθνής δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε. Πρέπει να βελτιωθούμε στον τομέα αυτό για να έχει η Ευρώπη πιο ισχυρή φωνή. Τα επόμενα πέντε χρόνια σαφώς και θα επιφέρουν αλλαγές. Στόχος μας θα πρέπει να είναι να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τους πόρους και να συμβλάβουμε υπόψη το κλίμα σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Θα είναι τιμή μου να συνεργαστώ μαζί σας και με το Κολέγιο των Επιτρόπων για να εξασφαλίσουμε ότι η αυριανή Ευρώπη είναι πιο βιώσιμη από τη σημερινή. Σας ευχαριστώ. Uh, thank you Ευχαριστούμε πολύ κυρία Χέντεγκαρτ για την παρουσίασή σας. Είσαστε η πρώτη υποψήφια που κράτησε ο λόγος της ο εισαγωγικός ακριβώς με ακρίβεια δευτερολέπτου 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα και σας ευχαριστώ και για τα μηνύματα που μας δώσατε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι η πιο φιλική προς το περιβάλλον περιοχή του κόσμου και πρέπει να μιλάμε με μια ενιαία φωνή στα θέματα αυτά. Ξεκινούμε την ακρόαση. Ξεκινούμε με τον Ρίχαρτ Ζέμπερ από το ΕΛΚ. Καλημέρα σας κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καλημέρα κυρία Υποψήφια Επίτροπε. Έχετε, σας εύχομαι κάθε τύχη γιατί έχετε να αναλάβετε ένα από τα πιο δύσκολα χαρτοφυλάκια και φυσικά έχετε την ε, εμπειρία στον τομέα αυτό και όπως είπατε ήδη στην ε, ε, παρέμβασή σας στην εισαγωγική είναι μια κλασική εγκάσια αρμοδιότητα η κλιματική αλλαγή η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί περαιτέρω και σε παγκόσμιο επίπεδο. Εγώ θέλω να, να, σας ε, θέσω ορισμένα ερωτήματα. Αναφέρατε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε την, τους ανταγωνιστές μας την Κίνα η οποία παράγει ανεμογεννήτριες πιο πολύ από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο, οι Αμερικανοί οι οποίοι λαμβάνουν άλλα μέτρα Πώς, κατά την άποψή σας λοιπόν, θα πρέπει να αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς θα πρέπει να προχωρήσει σε συγκεκριμένα επίπεδα πολιτικής, ποια εργαλεία θα πρέπει να εφαρμόσει μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, πώς θα είμαστε σε διαφορετική κατάσταση μετά από πέντε χρόνια. Ευχαριστώ. Έχουμε θέσει τους στόχους μας για τις ανανεώσιμες ενέργειες, Θέλουμε να είμαστε ενεργειακά αποδοτικοί. Έχουμε το στόχο για τη μείωση των εκπομπών. Νομίζω ότι οι στόχοι υπάρχουν. Η πρόκληση τώρα όμως για τα επόμενα πέντε χρόνια θα είναι να εφαρμόσουμε αυτούς τους στόχους. Όπως είπα υπάρχουν τομείς όπου μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Σε εθνικό επίπεδο δουλεύουμε για τον επιμερισμό των προσπαθειών. Υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες. <clears throat> Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν ε, Τομεί όπως όπου Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Παραδείγματος χάρη μεταφορές, όπως ανέφερα. Υπάρχουν πολλές ε, προτάσεις ε, που θα πρέπει να κάνουμε τα επόμενα χρόνια για τα φορτηγά, αλλά υπάρχουν και άλλοι τομείς ε, στις μεταφορές που μπορούμε να ασχοληθούμε. Παραδείγματος χάρη, ένα άλλο τομέα είναι η ναυσιπλοεία. Θα ήθελα να υπάρχουν διεθνείς κανόνες για την ναυσιπλοεία. Ελπίζω να είναι τμήμα της Συμφωνίας Κοπενχάγη. Η Ευρώπη θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα επόμενα χρόνια με κάποιο τρόπο θα αντιμετωπίσουμε και τις εκπομπές ε, από τα πλοία. Στα πλαίσια διεθνών κανόνων. Όταν ε, διαμορφώσουμε τις αγροτικές μας πολιτικές, επίσης θα πρέπει να ενσωματώσουμε νέες τεχνολογίες ούτως ώστε να είμαστε πιο κλιματικά φιλικοί ε, σε ό,τι αφορά την παραγωγή τροφίμων, ε, τις καλλιέργειες. Και επίσης θα πρέπει να είμαστε έξυπνοι. Όχι μόνο στην κατασκευή νέων κτηρίων, έχουμε ήδη πρωτοβουλίες, αλλά όταν ανακαινίζουμε, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι το κάνουμε το καλύτερο δυνατό τρόπο για τις επόμενες γενιές. Δεν μιλάω για το χρονικό ορίζοντα 2020 μόνο, αλλά και για το χρονικό ορίζοντα το μακρύτερο, 2050. Έχετε αναφέρει ορισμένα θέματα εφαρμογής τα οποία προήλθαν από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κοπεχάγη που δεν έγιναν δεκτά από άλλα κράτη-μέλη όμως, από άλλες χώρες μάλλον του κόσμου. Θεωρείτε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να επεκτείνει αυτά τα μέτρα και να τα εφαρμόσει και να πείσει όλα τα κράτη-μέλη να επεκτείνουν και σε άλλους τομείς τα μέτρα αυτά και με ποιο τρόπο από τη δική σας πλευρά εσείς θα δράσετε ώστε να γίνει αυτό σε συγκεκριμένο επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι υπάρχει μία πρόκληση. Αφενό να θέσουμε του στόχου, αλλά αφετέρου να έχουμε και τα εργαλεία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν 3.000 διαφορετικές ε, περιπτώσεις όπου τα κράτη-μέλη δεν κάνουν αυτό που θα έπρεπε να κάνουν. Σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να προχωρήσουμε. Ε, αυτά είναι γενικά λόγια βέβαια. Γιατί στο επίπεδο του κλίματος υπάρχουν ε, συγκεκριμένα εργαλεία για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την έλλειψη της εφαρμογής. Παραδείγματο χάρη, αν δεν εφαρμόζεται τις καθορισμένες κλιματικές πολιτικές με βάση το Κιώτο. Υπάρχουν διεθνείς κανόνε όπου μπορείτε να, ε, μπορεί να σας επιβληθεί πρόστιμο. Υπάρχουν τρόποι για να εξασφαλίσουμε την εφαρμογή. Αλλιώς θα, πληρώσετε αν δεν το κάνετε. Ή θα πρέπει ας πούμε να παραχωρήσετε τα δικαιώματά σας. Αν στην πρώτη περίοδο αυτό που έπρεπε να κάνετε δεν το κάνετε. Θα πρέπει μετά ας πούμε να υπάρχει ένα τίμημα για σας. Will η επόμενη ερώτηση. Η σύνοδος Κορυφή τη Κοπεχάγης ήταν, απο... η σύνοδος ήταν αποτυχία και ήσασταν τμήμα αυτή τη συνόδου. Ήσασταν ε, από τους ανθρώπους που είχαν ε, ένα ρόλο κλειδί σε αυτή τη σύνοδο. Η ΕΠΑ και η Κίνα ε, πίεζαν τα πράγματα, ενώ εμείς ήμασταν απόντες. Τι πρωτοβουλίες θα λάβετε αν γίνετε δεκτή ως Επίτροπος, ούτω ώστε να αποκτήσουμε εκ νέου αυτόν τον ηγετικό ρόλο για την καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή. Δεν μιλάω μόνο για την εφαρμογή, αλλά και για νέε πρωτοβουλίε. Όταν, παραδείγματο χάρη, πότε θα προτείνετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξήσει τι δεσμεύσει τη για τη μείωση των εκπομπών από το 20% στο 30%. Καταρχά, όπω είπα και προηγουμένω, θα ήθελα να είχαμε προχωρήσει περισσότερο στην Κοπενχάγη. Αλλά μην ξεχνάμε ότι Μιλήσαμε για τη χρηματοδότηση και όλες οι αναπτυσσόμενες οικονομίες ε, δέχονται ότι έχουν ε, ευθύνη και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Και πριν την Κοπενχάγη, εξαιτία του γεγονότος ότι είχαμε θέσει αυτή την προθεσμία πριν από τρία χρόνια, η Βραζιλία, η Νότια Αφρική, η Ινδία, η Κίνα και οι Ηνωμένε Πολιτείε, όλε οι χώρε που δεν ήταν τμήμα της, του πακέτου του Κιώτο, έθεσαν στα εθνικά του συστήματα προ, προτάσεις και στόχους για να δράσουν σε εθνικό επίπεδο. Επομένω, νομίζω ότι κάτι κάναμε, ουσιαστικό μάλιστα, στην Κοπενχάγη. Επίσης, πετύχαμε το στόχο του, των δύο βαθμών Κελσίου. Όπως είπα στην πρώτη μου παρουσίαση, βέβαια, δεν τα έχουμε καταφέρει όλα. Είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει τον ηγετικό ρόλο. Ε, Απλώ θέλω να τονίσω ότι πρέπει να είμαστε πιο ενωμένοι, να μιλάμε μια φωνή. Ε, φυσικά εύκολα να το λέει κανεί, πάνω να το κάνει. Αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε τι, έγιναν, ε, τι έγινε τις τελευταίες 24 ώρες στην Κοπενχάγη. Γιατί στα διεθνή βήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι πιο ενωμένη αν θέλει να ακουστεί. Ένα τομέα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα μπορούσε να είχε παίξει πιο σημαντικό ρόλο θα ήταν αν είχε κάνει προσφορές χρηματικές νωρίτερα. Πολύ αργά ήρθαν αυτέ οι προσφορέ, Πολύ αργά φτάσαν στο τραπέζι. Νομίζω ότι αν είχε γίνει νωρίτερα αυτό θα είχε θετικό αντίκτυπο στι αναπτυσσόμενες χώρε. Αν πριν να φύγουν από τι πρωτεύωσέ του, οι αξιωματούχοι είχαν δει ότι φτάνουν τα κονδύλια θα είχαν αλλάξει στάση. Ε, σε ό,τι αφορά το 30% εγώ θέλω να πετύχουμε το 30% το συντομότερο δυνατό. Αλλά εκ των υστέρων βλέποντα αυτά που έγιναν στην Κοπενχάγη θεωρώ ότι θα πρέπει μέχρι την 1η ε, Φεβρουαρίου θα πρέπει να μην ζητήσουμε έτσι αστόχαστα το, α, την μετάβαση από το 20% στο 30%. Ευχαριστώ για την απάντησή σας. Τώρα, για τη χρηματοδότηση και το πόσο σημαντική είναι. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Έχετε ένα μικρό χαρτοφυλάκιο και θα πρέπει να δουλέψετε πολύ ε, και να συνεργαστείτε πολύ στενά και να συμφωνήσετε με άλλους επιτρόπους. Ε, φτάνετε στην, στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα χαρτοφυλάκιο που δεν έχει πολλά χρήματα. Τι θα κάνετε. Ε, μιλήσατε για τη γεωργία ήδη στην εισαγωγή σας. Ε, θα προσπαθήσετε να κερδίσετε κάποια κονδύλια από τον γεωργικό προϋπολογισμό. Ξέρω πολύ καλά ότι δεν κολυμπάμε στο χρήμα. Ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, <laughs> ούτε στα κράτη-μέλη ε, ζούμε σε παχέ αγελάδε. σωστό είναι αυτό που περιγράψατε. Όταν ε, μιλήσουμε για τις ε, δημοσιονομικές προοπτικές, είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε καλύτερο συντονισμό ανάμεσα σε αυτό που λέμε ότι είναι οι πολιτικές μας προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο και σε αυτό που καταστούμε ως προτεραιότητα στον προπολογισμό μας. Νομίζω ότι πολλά θα κερδίσουμε αν πρασινίσουμε εντό αγωγικών τη γεωργία μας. Αν επενδύσουμε σε νέες τεχνολογίες, αν κάνουμε προγράμματα επίδειξης στον γεωργικό τομέα, μπορούμε να εκμοντερνίσουμε τη γεωργία με έναν τρόπο όχι μόνο θα είναι πιο φιλοπεριβαλλοντικός, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να εξάγουμε αυτή την τεχνογνωσία ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, είναι μια τεράστια πρόκληση το πώς θα καταστεί πιο φιλική για το περιβάλλον η Γεωργία. Ακολουθεί ο Κρίς <clears throat> Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, σας βλέπω σαν μια δυναμική υπουργό ε, περιβάλλοντος και ήταν πάρα πολύ ευχάριστη τις προηγούμενες συζητήσεις μας, ακόμα και αν δεν συμφωνούσαμε πάντα. Όταν ανακοινώθηκε ότι προτείνεστε εσείς ως ε, ε, επίτροπος κλιματικής δράση σκέφτηκα είναι ένας ρόλος που σας πηγαίνει τέλεια. Αλλά τα πρότυπα που έχει θέσει τον εαυτό τη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Κοπεχάγη οδήγησαν σε μια αποτυχία. Δεν πλησιάσαμε καν σε αυτά τα πρότυπα τα οποία θέλαμε να έχουμε. Και τώρα, γιατί θέλουμε να έχουμε ένα ε, επίτροπο για κλιματική δράση μετά από μια τέτοια αποτυχία. Σα ευχαριστώ για το ερώτημα αυτό. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό να μπορώ να το απαντήσω εδώ και να μην κάνω απλώ συζητήσει στου διαδρόμου. Μπορεί να επικρίνει κανείς πάρα πολύ αυτά τα οποία έγιναν στην Κοπενχάγη, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι δίκαιο να επικρίνει κανείς αυτούς οι οποίοι δαπάνησαν χρόνια για να προσπαθήσουν να κινητοποιήσουν τον κόσμο στον πλανήτη μας. Δεν πετύχαμε ακριβώ αυτό το οποίο θα θέλαμε να έχουμε. Αυτό που θα θέλατε εσεί να πετύχετε, αυτό που θα θέλαμε εγώ να πετύχω στην Κοπενχάγη. Αλλά όπω είπα στην αρχή, ποιο θα είχε φανταστεί πριν από μερικά μονάχα χρόνια ότι μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν να πείσουμε όλες τις αναδυόμενες οικονομίες να αποδεχθούν ότι είναι συνυπεύθυνες για την κλιματική αλλαγή. Αυτή ήταν η επιτυχία της Κοπενχάγης. Ναι, οι αναπτυγμένες χώρες δεν μπορούσαν να καταλήξουν σε δεσμεύσεις να μειώσουν τις εκπομπές τους, αλλά οι αναδυόμενες οικονομίες δέχτηκαν ότι πρέπει και αυτές να συμμετάσχουν στην κοινή αυτή δράση. Και αυτό γίνεται όχι μόνο σε διεθνέ επίπεδο, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Δέχονται ότι πρέπει να έχουν ανακοινώσει για τα θέματα αυτά και την πρόοδο που επιτυγχάνεται. Νομίζω ότι έχουμε πετύχει πολλά. Και στην προσέγγιση <clears throat> τη διάσκεψη Κοπεχάγη είχαμε τονίσει ότι αν θα θέταμε μεγάλη πίεση στου εταίρου μα, θα έπρεπε να προετοιμαστούν καλύτερα για να έρθουν στην Κοπεχάγη. Τελικά απέδωσε αυτή η στρατηγική. Για κάποιου λόγου, ορισμένε χώρε αποφάσισαν την τελευταία στιγμή ότι δεν θα ήθελαν να δεσμευτούν για, συγκεκριμένα, για συγκεκριμένους στόχους. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το επιρρύψει κανείς στη Δανική Προεδρία ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήταν κρίμα να κατηγορήσουμε αυτούς οι οποίοι δραστηριοποιήθηκαν περισσότερο από οποιουσδήποτε άλλους για να τροποποιήσουν την διεθνή νοοτροπία για τα θέματα αυτά λόγω της αντίδρασης αυτών οι οποίοι δεν θέλησαν να προχωρήσουν. Ευχαριστώ. Και πάλι σας λέω ότι σας βλέπω ότι έχετε πολύ ενθουσιασμό και πολύ, <laughs> πολύ ενδιαφέρον για το χαρτοφυλάκιό σας. Όλοι μας θέλουμε να έχουμε, πολλοί από εμάς θέλουμε να έχουμε ένα πραγματικά καλό επίτροπο ο οποίος θα προχωρήσει στα θέματα αυτά και θα πιέσει μέσα στο Σώμα των Επιτρόπων. Ένα μεγάλο μέρος του έργου σας θα καλύπτει και την ε, Κομισιόν, αλλά θα πρέπει να ε, είσαστε σε επαφή με το Συμβούλιο. Πού νομίζετε ότι βρίσκεται η ισορροπία μεταξύ του να είσαστε μαχητικοί από τη μια μεριά και αδιάλακτοι και του να είσαστε συνδιαλλακτικοί και να συνεργάζεστε με τους άλλους. Δεν μπορώ να καθορίσω μια συγκεκριμένη οριοθετική γραμμή γιατί αυτό το οποίο είναι σωστή ισορροπία για ορισμένους δεν είναι η σωστή ισορροπία για άλλους. Αλλά η πολιτική φυσικά σημαίνει ότι πρέπει να τολμάει κανείς να αγωνίζεται για τα πράγματα τα οποία πιστεύει. Ορισμένε φορές έχετε μάχε, έχετε να αντιμετωπίσετε μάχε. Αλλά άμα δεν θέλει κανεί να δίνει μάχε, δεν πρέπει να είναι μέσα στην πολιτική. Είναι σημαντικό να τροποποιήσουμε το υπόδειγμα τη κοινωνία μα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε σε επίπεδο απασχόληση, χρήση ενέργεια, όλα αυτά τα θέματα τα οποία διακυβεύονται στην ε, Κοπεχάη και στην κλιματική αλλαγή. Τότε θα πρέπει να υπάρξουν μάχε για όλα αυτά τα θέματα όταν δεν υπάρχει ομοφωνία και πρέπει κανεί να είναι δυναμικό. Η Κομισιόν δεν είναι μονάχα σε μια κυβέρνηση πρέπει πολλές φορές να λειτουργεί κανείς και μέσα από τους συναδέλφους στην Κομισιόν. Αλλά νομίζω ότι όλο και περισσότερο η Ευρώπη θα κατανοήσει ότι αν δεν προχωρήσουμε μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, εάν δεν εφαρμόσουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε υποσχεθεί, τότε τελικά θα υπολοιπόμεθα τον άλλον και θα χάσουμε όχι μόνο σε επίπεδο περιβάλλοντο, αλλά θα χάσουμε και σε επίπεδο απασχόληση και αυτή η αναγνώριση νομίζω ότι είναι όλο και πιο διαδεδομένη ακόμα και στου βιομηχανικού κύκλου. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό αξίζει τον κόπο να το προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Η του χάσει. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, μου άρεσε η δήλωσή σας ότι θέλετε η Ευρώπη να είναι η πιο περιβαλλοντικά φιλική περιοχή του κόσμου. Είστε έτοιμοι να είστε επίσης σκληροί και έναντι της πιο ε, ρηπαίνουσας μορφής παραγωγής ενέργειας, παραγωγή με άνθρακα, γιατί το υφιστάμενο σύστημα εμπορίας εκπομπών δεν αρκεί για να αλλάξουν τα πράγματα. Βλέπουμε ακόμα να κατασκευάζονται ε, μονάδες άνθρακα θα θεσπίσετε κανόνες για να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρξει μετάβαση μακριά από τον μονάδες άνθρακα και τουλάχιστον θα κάνετε μελέτες αντικτύπου εντός ενός έτους. Απάντηση. Κατανοώ το ερώτημά σας. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι όταν μιλάμε για μονάδες παραγωγής με άνθρακα είναι τμήμα του συστήματος εμπορίας εκπομπών μπορούμε να έχουμε και πρότυπα επιδόσεων και στη γραπτή απάνταση θα σας είπα ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε το εάν η τεχνολογία αυτή δουλεύει πριν αλλάξουμε τα πράγματα. Νομίζω λοιπόν ότι δεν θα πρέπει να βιαστούμε και επίσης πιστεύω ότι αν έχουμε τέτοιου είδους πρότυπα επιδόσεων για τις νέες μονάδες, πώς θα έχουμε την εγγύηση ότι κάποιες χώρες δεν θα παρατείνουν απλώς τη διάρκεια ζωής των παλαιών μονάδων και πιστεύουμε ότι προβλέπουμε ότι θα κατασκευαστούν περίπου 60 μονάδες παραγωγής ενέργειας για τα επόμενα 60 χρόνια και καθώς κάποια κράτη-μέλη και νέα κράτη-μέλη δεν θα έχουν ελεύθερη δωρεάν ε, παροχή εκπομπών για αυτές τις νέες μονάδες ενώ θα έχουν για τις παλιές. Να μην ενθαρρύνουμε λοιπόν τα κράτη-μέλη να διατηρήσουν σε λειτουργία τις παλαιές μονάδες, γιατί σε πολλές περιπτώσεις είναι καλό να ε, εφαρμοστεί η νέα τεχνολογία. Διστάζω λοιπόν να σας το υποσχεθώ αυτό, γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε το εάν η τεχνολογία αυτή ε, δουλεύει και επίσης χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για να τα εξοπλίσετε. Αν έχετε τρεις μονάδες απαιτείται η ενέργεια ισοδύναμη με τέσσερις μονάδες για να τα εξοπλίσετε και με την διαδικασία δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα. Συμπληρωματική απάντηση, ερώτηση, συγγνώμη. Καταλαβαίνω, δεν θέλετε να βιαστείτε, αλλά δεν είπατε Κάνω ότι δέχεστε να κάνετε μία μελέτη αντικτύπου. οι Τα πρότυπα αποδόσεων μπορούν να εξαρτηθούν και από την ηλικία της μονάδας. Αν διστάζετε λοιπόν τόσο πολύ για αυτό το θέμα και ταυτόχρονα μιλάτε για στόχους μείων 30%. Αλλά αν όμως καθυστερήσετε την απόφαση να δεσμευτούμε για μείον 30% στις εκπομπές, τι μέτρα θα λάβετε για να εξασφαλιστεί ότι θα το κάνουμε με, θα, επιτύχουμε τους στόχους αυτούς με κάποια τρίκ να προσμετρήσουμε δάσεις στα αναπτυσσόμενες χώρες παραδείγματος χάρη. Απάντηση. Δεν είπα ακριβώς αυτό. Είπα ότι εάν τελικά λάβουμε αυτή την απόφαση πρέπει να την ξανασκεφτούμε γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποιες αρνητικές παρενέργειες που δεν θα θέλαμε να τις δούμε και βεβαίω με μια μελέτη αντικτύπου θα μπορούσαμε να αξιολογήσουμε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Απλώ λέω ότι είναι ένα θέμα που δεν είναι άσπρο ή μαύρο και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να μην είμαστε, να επιβάλλουμε υπερβολική ρύθμιση σε οποιοδήποτε τομέα. Κύριος Μάρτιν Κάλαχαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με την έγκριση του πακέτου για την κλιματική αλλαγή το Δεκέμβριο του 2008 η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε σε ανταγωνιστικά μειονεκτική θέση την βαριά της βιομηχανία έναντι άλλων χωρών. Τη βιομηχανία που χρησιμοποιεί εντατικά την ενέργεια. Και αυτό θα παραμείνει μέχρι ότου οι εταίροι μας και οι αναπτυσσόμενες χώρες συμφωνήσουν να υπάρχουν δεσμευτικά μέτρα, τα οποία φυσικά θα πρέπει να δεσμεύουν ε, τις ΗΠΑ, Κίνα, Ινδία και τις υπόλοιπες χώρες σε κοινή δράση μαζί μας. Εάν όχι όμως, αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, πώς θα μπορέσετε να μετριάσετε τα ανταγωνιστικά προβλήματα τα οποία προκύπτουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να πείσετε τις αναπτυσσόμενες χώρες και τις άλλες χώρες να κάνουν κάτι. Σίγουρα υπάρχει ο κίνδυνο τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων, τη λεγόμενη διαρροή άνθρακο. Ό,τι και να κάνουμε στον τομέα αυτό θα πρέπει να βασίζεται σε μια ισορροπία. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να είμαστε υπερβολικά ισορροπημένοι, τόσο υπερβολικά ισορροπημένη και επιφλακτική ότι τελικά δεν θα αποκομίσουμε κανένα όφελος. Όπως είπα στην αρχή, πιστεύω ότι είτε πετύχουμε διεθνή συμφωνία ή όχι, η Κίνα προχωράει με, με, γρήγορα βήματα. Πέρσι η Κίνα ήταν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ηλιακής, ε, ηλιακών συλλεκτών, φέτος είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ε, ανεμογεννητριών. Αυτό δείχνει λοιπόν ποια είναι η πραγματικότητα. Ξέρω ότι οι βιομηχανίες δεν θέλουν ρυθμιστικές, ε, ρυθμιστικούς περιορισμούς και λένε δεν μπορούμε να το κάνουμε, μη μας πιέζετε τόσο πολύ, θα μας φάνει οι ανταγωνιστές μας κτλ. Αλλά βλέπουμε ότι τα πράγματα αλλάζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλάζουν στην Κίνα, αλλάζουν στην Ινδία. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί δεν πρέπει για λόγους καλών προθέσεων να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τις δικές μας βιομηχανίε. και με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά θα τις κάνουμε να χάσουν το παιχνίδι, να χάσουν το μερίδιο της αγοράς του εν καιρό. Πρέπει να εξισορροπήσουμε φυσικά όλα αυτά, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε τόσο φιλικοί μέσα σε εισαγωγικά στις βιομηχανίες μας, ώστε να μην τους επιτρέψουμε να ανανεωθούν και να είναι ανταγωνιστικές στο μέλλον. Γιατί πιστεύω ότι πρέπει να σπρώξουμε απαλά αλλά αποφασιστικά την ευρωπαϊκή βιομηχανία στη σωστή κατεύθυνση. Όχι λόγω αυτού που γίνεται στην Κίνα, στις Ηνωμένε Πολιτείε ή αλλού, αλλά γιατί το απαιτεί η Ευρώπη για να μπορέσει να προστατεύσει το περιβάλλον της και το κλίμα του πλανήτη μας. Δεν είμαι εναντίον του να σπρώχουμε τη βιομηχανία προς τη σωστή κατεύθυνση. Σίγουρα <clears throat> η Κίνα έχει προχωρήσει πολύ στην πράσινη τεχνολογία, αλλά έχει και μεγάλο αριθμό ε, σταθμών ενέργειας που χρησιμοποιούν άθρακα. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε και τα δύο. Γιατί απλώς να δεχτούμε να μεταφερθούν όλες οι βιομηχανίες οι οποίες είναι μεγάλης έντασης ενέργειας μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτό συμβαίνει τελικά. Δεν είναι ένα παιχνίδι που γίνεται ή το ένα ή το άλλο. Μπορούμε να προωθήσουμε τις πράσινες ε, τεχνολογίες, αλλά εάν δεν υπάρξει δέσμευση από την Κίνα και τις ε, άλλες αναπτυσσόμενες χώρες θα προχωρήσουν σε παραγωγή νέων τεχνολογιών αλλά θα απορροφήσουν και τις βιομηχανίες που εμείς διώχνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ μαζί σας. Γι' αυτό εδώ και χρόνια εργάζομαι προσπαθώντας να πείσω την Κίνα και άλλες αναδυόμενες οικονομίες να συμφωνήσουν μαζί μας σε ένα διεθνές καθεστώς για το κλίμα και την κλιματική αλλαγή. Αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να πράξουμε. Γιατί για πολλούς λόγους και άμα το δούμε από ευρωπαϊκή οπτική γωνία και βάσει της ανάλυσης που μας δώσατε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα να ρηπαίνουν δωρεάν οι αναπτυσσόμενες οικονομίες, οι αναδυόμενες οικονομίες. Γι' αυτό νομίζω ότι η Κομπεχά ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Η επόμενη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι τι θα γίνει την 1η Φεβρουαρίου. Θα διεθνοποιήσει πράγματι η Κίνα του στόχους που ενέκρινε εσωτερικά, σε εθνικό επίπεδο. Αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις επερχόμενες <clears throat> κλιματικές διαπραγματεύσεις και για την προοπτική να δεχθεί και ένα κάποιο διεθνές καθεστώς, το οποίο φυσικά θα είναι και προς το συμφέρον των δικών μας βιομηχανιών. Καρτίκα Λιωτάρ, η επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ. Και καλώς ήρθατε κυρία Χέντεγκάρντ. Ένας από τους βασικούς στόχους για να, και για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή είναι για να έχουμε ένα πιο φιλοπεριβαλλοντικό ενεργειακό μείγμα. Είπατε ότι στις απαντήσεις σας ότι η πυρηνική ενέργεια θα είναι βασικό τμήμα αυτού του μείγματος. Εγώ νομίζω ότι η πυρηνική ενέργεια είναι οτιδήποτε άλλο παρά βιώσιμη. Και πριν από τη συνάντηση της COP15, όταν συναντηθήκαμε με την Επιτροπή, ε, μάθαμε και καταλάβαμε ότι τελικά η Επιτροπή δεν είχε καμία θέση. Τώρα, ποια είναι, αυτή, ποια είναι η άποψή σας για αυτή τη στάση της Επιτροπής, ότι δεν έχουμε άποψη δηλαδή. Και ποια είναι η προσωπική σας θέση για την πυρηνική ενέργεια και τη βιωσιμότητα. Νομίζω ότι εδώ και καιρό η ευρωπαϊκή πολιτική ήταν ότι το ενεργειακό μείγμα αποφασίζεται από τις ίδιες τις χώρες. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα όπου αποφασίσαμε με ψήφο ε, στο Κοινοβούλιο το 85 ότι δεν θέλουμε πυρηνική ενέργεια και αποφασίσαμε ότι θα προχωρήσουμε με τις ανανεώσιμες, με την ενεργειακή αποδοτικότητα και τα καταφέραμε περίφημα. Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο εγώ μεγάλωσα και λειτουργήσα. Αλλά η πυρηνική ενέργεια υπάρχει στον κόσμο και θα υπάρχει τα επόμενα χρόνια, για πολλά χρόνια. Είναι πραγματικότητα λοιπόν. Και γι' αυτό είναι σημαντικό είναι να εξετάσουμε τα θέματα ασφάλειας της πυρηνικής ενέργειας. Γι' αυτό η Euratom και άλλα θεσμικά όργανα και οργανώσεις με την τεχνολογία και την ανάπτυξη σε αυτόν τον τομέα προσπαθούν ε, να εξασφαλίσουν ότι οι πυρηνικοί αντιδραστήρες που υπάρχουν είναι όσο δυνατόν πιο ασφαλείς. Στο δικό μου μυαλό πάντως η πυρηνική ενέργεια δεν είναι σε καμία περίπτωση ανανεώσιμη και βιώσιμη μορφή ενέργειας. Ωραία. Πέρα από το ενεργειακό μείγμα, υπάρχουν και άλλες δράσεις που θα προωθήσετε για να καταπολεμήσετε την κλιματική αλλαγή. Η επόμενη λοιπόν ερώτησή μου είναι, αν θα προωθήσετε δράσεις για τις εκπομπές του μεθανίου, που είναι ένα τεράστιο και πολύ σημαντικό αέριο. Τι θα κάνετε με αυτό το θέμα. Θα ενθαρρύνετε επίσης τον κόσμο να τρώει ε, τρόφιμα τα οποία παράγονται τοπικά, ούτως ώστε να μειωθούν οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα. Ε, και να μην τα φέρνουμε από την άλλη μεριά του πλανήτη. Καλύπτεται ένα πολύ ευρύ ε, πεδίο. Επιστητούμε το ερώτημά σας. Κανονικά πρέπει το συμπληρωματικό σας ερώτημα να αναφέρεται στο προηγούμενο ερώτημα. Στις διεθνείς διαπραγματεύσεις θα πρέπει να δούμε αν οι πιο επικίνδυνες ουσίες θα πρέπει να συμπεριληφθούν. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε και στην Κοπενχάγη. Τώρα, το θέμα για τις, ε, τα τρόφιμα που παράγονται τοπικά Μακάρι. Μακάρι να καταλάβει ο κόσμος ότι έχει νόημα και για λόγους κλιματικούς να αγοράζουν πράγματα τα οποία παράγονται κοντά ή που είναι εποχιακά τρόφιμα. Αλλά σε μια παγκόσμια οικονομία θα πρέπει να ρυθμίζουμε πολιτικά με διαφορετικά, διαφορετικό τρόπο αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει ο καθένας να έχει και επιλογές, αλλά θα πρέπει οι, οι εκπομπές από τα πλοία, από τα αεροπλάνα να συμπεριλαμβάνονται. Αν λοιπόν ε, εσύ τρως τρόφιμα τα οποία εισάγονται από πολύ μακριά, θα πρέπει κάπως να πληρώνεις το τίμημα. Και με αυτόν τον τρόπο υπάρχει ε, ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για τα τρόφιμα που παράγονται και καταναλώνονται τελικά τοπικά. Η Άννα Ρόσπαχ το επόμενο ερώτημα. Ευχαριστώ κυρία Χάντεγκάρτ. Ε, σας ευχαριστώ για την ενημέρωση που κάνετε σε αυτήν την Επιτροπή κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της COP15. Δεν είναι καθόλου α, καταφρονητέα η προσπάθεια που κάναμε για να συγκεντρώσουμε όλους τους αρχηγούς α, κρατών και κυβερνήσεων ε, σε ένα τόπο. Ξέρετε τώρα για τον Off ότι οι εστονικές οργανώσεις πήγαν την ε, Γερμανία και... και τη Φιλανδία και τη Γερμανία στο δικαστήριο. Τι θα γίνει ε, με τα απόβλητα που φτάνουν στην Ευρώπη από διάφορες μονάδες παραγωγής ε, ηλεκτρικής ενέργειας. Καταρχάς γνωρίζω ότι διάφορες ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις ανησυχούν πάρα πολύ για, για τον ε, αγωγό North Stream φυσικού αερίου. Θα πρέπει να γίνει μια μελέτη αντικτύπου σε εθνικό επίπεδο και θα πρέπει να δούμε τι θα πρέπει να κάνουμε με το περιβάλλον. Γνωρίζω αυτό το θέμα ε, από Δανέζικη Σκοπιάς. Και αν δείτε και πώς είναι και η θάλασσα εκεί, θα πρέπει να δούμε αν ε, πρέπει να δώσουμε άδεια για ένα τέτοιο project ε, το οποίο θα περνάει από τη θάλασσα. θα πρέπει να πληρούνται διάφορα περιβαλλοντικά κριτήρια. Οι Σουηδοί και οι Φιλανδοί επίσης πρέπει να κάνουν παρόμοιες αναλύσεις. Και θα πρέπει να έχουμε μια συνολική προσέγγιση. Και μόνο ε, αν τα περιβαλλοντικά πρότυπα τηρούνται, τότε μόνο θα πρέπει να πάρει το πράσινο φως ε, το Nord Stream. Υπάρχει τώρα και μια πιο πολιτική διάσταση. Είπατε ότι θα πρέπει να γίνουμε ανεξάρτητοι ενεργειακά. Υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις, ανεξάρτητα από τη Ρωσία. ναι, μεν είμαστε εξαρτημένοι στην ε, Ευρώπη από τη Ρωσία και από το φυσικό της αέριο, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε γιατί θέλουμε τον αγωγό. Μήπως είναι καλύτερο να έχουμε πολλαπλούς ε, αγωγούς παρά να έχουμε έναν ή πολύ λίγους. Γι' αυτό λοιπόν το σκέφτηκε η Ευρώπη, μήπως θα πρέπει να έχει περισσότερους αγωγούς ευθύς εξ αρχής. Και αν μπορούμε να φτιάξουμε αυτούς τους αγωγούς με βάση το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, θα πρέπει να το δούμε αυτό. Συμπληρωματική ερώτηση. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι όταν το εξετάζουμε αυτό το θέμα, Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν πολλές βόμβες ε, στο βυθό της θάλασσας ε, που δεν έχουν ε, εκραγεί από τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αν έρθει σε επαφή η βόμβα με τον αγωγό, τι γίνεται. Επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα είναι τι γίνεται με τα απόβλητα από το, το δίκτυο διανομής της ενέργειας που, είναι, που έχει παλιώσει. Απάντηση. Όντως υπάρχει τέτοιο πρόβλημα με βόμβες που δεν έχουν εκραγεί. Ξέρουμε όμως που βρίσκονται αυτές οι βόμβες και μπορούμε να αλλάξουμε το... την πορεία του αγωγού. Φυσικά δεν έχουν τελειώσει οι έρευνες. Οι φιλανδικές και οι σουηδικές ε, αρχές θα κάνουν και αυτές ε, έλεγχο. Πάντω η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει μια γενική εποπτεία και θα δώσει το πράσινο φως μόνο εφόσον όλα τα τμήματα της αλυσίδα λειτουργούν όπως πρέπει. Ευχαριστώ κυρία Ρόσπαχ. Σίγουρα όλοι ξέρουν ότι δεν υπάρχει πια συνωμοσία, αλλά αυτόν που θέλουν να κάνουν να πιστεύουμε ότι αλλάζει το κλίμα. Ξέρουμε όλοι ότι δεν υπάρχει καθόλου αμφισβήτηση για την κλιματική αλλαγή. Επομένως δεν υπάρχει το πρόσθετο αυτό ερώτημα το οποίο περιμένατε να βρεθεί. Ερχόμαστε τώρα στη δεύτερη φάση των ερωτήσεων. Ξεκινάμε με τον Καλ Χάιτ Φλόρεν. Είναι κρίμα που δεν είναι εδώ οι αρνητέ τη κλιματική αλλαγή για να μπορέσουμε να, συζητήσουμε, να συζητήσουμε μαζί του. Θα ήθελα να πω κάτι σε σχέση με αυτά που είπε ο φιλελεύθερο φίλο μα, ο Κρι Ντέβι, την πρώτη εβδομάδα στην Κοπεχάγη. Ήταν παρόν και εκεί ήταν όλοι οι γραφειοκράτε και επομένω δεν έγινε κάτι το ιδιαίτερα έντονο. Όταν ήταν όμω κοινοβουλευτικοί παρόντε ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα και αντιμετωπίσανε φυσικά τον τρόπο λειτουργία των Κινέζων, ο οποίο ήταν ιδιαίτερα δραματικό. Κυρία Επίτροπε, υποψήφια Επίτροπε, έχω ακούσει πολλά πράγματα για τη φιλοσοφία που ακολουθείτε. Εγώ πιστεύω ότι η πολιτική σας να έχετε μια αυστηρή πολιτική κυρώσεων στην Ευρώπη ήταν επιτυχής. Πώς θα μπορούσαμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε να γίνει η κλιματική αλλαγή από πρόβλημα σε μια δυνατότητα να μιλήσουμε για μεγαλύτερη αποδοτικότητα, επομένω μεγαλύτερες εξαγωγικές δυνατότητες, μεγαλύτερη ασφάλεια τροφοδοσίας με ε, πρώτες ύλες. Πώς λοιπόν μπορούμε να, το, να αυξήσουμε αυτή τη συνειδητοποίηση μεταξύ του πληθυσμού. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν ακολουθήσαμε μια πολιτική κυρώσεων, μια πολιτική ποινικοποίηση στην ε, χώρα μου. Υπήρξαν κάποια πράγματα τα οποία χρειάστηκε να κάνουμε σε πολιτικό επίπεδο. Νομίζω όμως ότι είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να διευρύνουμε τον ορίζοντα αυτής της πολιτικής και εγώ θέλησα να τα πω αυτό και στην ε, αρχική μου παρουσίαση λέγοντας ότι η ατζέντα του κλίματος είναι και μια ατζέντα για δημιουργία θέσεων απασχόλησης, για να έχουν τα παιδιά μας καθαρότερο αέρα, καθαρότερα ύδατα. Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα από την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Είπα ότι σε ένα μέλλον όταν δεν θα υπάρχουν επαρκεί πόροι ή θα είναι σπάνιοι αυτοί οι πόροι, είναι οικονομικά απόλυτα λογικό και εύλογο να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε λιγότερους πόρου και λιγότερη ενέργεια. <clears throat> Ο η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας, ο Διεθνής Φορέας Ενέργειας, μας είχε, είχαμε έρθει σε επαφή μαζί τους και είπε ποια είναι η πορεία, ποια θα είναι η πορεία των ε, τιμών πετρελαίου. Εφόσον μειώνεται η παραγωγή θα ανέβουν και θα φτάσουν να είναι αστρονομικές εν καιρό οι τιμές του πετρελαίου. Πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε την προσοχή μας σε όλα αυτά τα θέματα. η Κοπενχάγη και η κινητοποίηση η οποία προεκλήθη στην Ευρώπη, θα πρέπει να έχει και ένα χαρακτήρα πιο ευχάριστο, να μπορούν τα, οι πολίτε να καταλαβαίνουν ποιε είναι οι ευκαιρίε, ποιε είναι οι δυνατότητε οι οποίε ανοίγονται. Εγώ είμαι από ένα συντηρητικό κόμμα στην Ευρώπη και ακολουθώ αυτή την ε, παράδοση, πιστεύω θα ήταν πολύ σημαντικό να αποφύγουμε μια κοινωνία που θα λέμε δεν θα κάνετε αυτό, αυτό απαγορεύεται, δεν έχετε καμιά επιλογή στο τάδε θέμα. Αυτό όμως σημαίνει ότι πρέπει να αντιδράσουμε έγκαιρα και όχι καθυστερημένα στην κλιματική αλλαγή. Όσο διστάζουμε, τόσο περισσότερο διακινδυνεύουμε να φτάσουμε σε μια πολιτική η οποία θα είναι κατασταλτική, αν θέλετε, για την κλιματική αλλαγή που δεν θα είναι αυτά τα εργαλεία τα οποία θα ήθελα και εγώ να χρησιμοποιήσω. Ευχαριστώ, δεν υπάρχει άλλο συμπληρωματικό ερώτημα. Ναι, ήταν πολύ σαφές, είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Ακολουθεί τώρα ο Ταν Γιόργενσεν. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και θα αναμένω από εσά μια πολύ αποδοτική συνεργασία εάν τελικά επιβεβαιωθείτε ως Επίτροπος. Αν δούμε την όλη όθηση που οδήγησε στην Κοπενχάγη και αν δούμε το πώς προσδιορίστηκαν οι διάφορες φιλοδοξίες, το τελικό αποτέλεσμα ήταν ένα φιάσκο, το οποίο ακόμα και εσείς προσεκτικά αναγνωρίσατε λέγοντας ότι θα μπορούσαμε να είχαμε και ένα πιο θετικό αποτέλεσμα. Εάν όμως τελικά θέλουμε η Ευρώπη να δώσει το παράδειγμα στην Ευρώπη, τότε θα πρέπει να είμαστε αρκετά ισχυροί για να μάθουμε από τα σφάλματά μας και να κάνουμε αυτοκριτική. Τα δύο πιο σοβαρά σφάλματα της Δανικής Προεδρίας για την Κοπενχάγη μπορείτε να τα σχολιάσετε παρακαλώ. Απάντηση είναι διατομιακή εμπειρία το να είμαι υπό το πυρ των ερωτήσεων σας εδώ. Αν καθορίσουμε προσδοκίες ή στόχους ε, πριν την Κοπενχάγη, αν είχαμε απλώς αφήσει τη διεθνή διαδικασία να προχωρά σιγά σιγά χωρίς να είχαμε βάλει κανένα χρονοδιάγραμμα, τότε πιστεύω και εσείς θα μπορούσατε επίσης να συμφωνήσετε κύριε Γιάννησεν ότι τα πράγματα θα είχαν τελικά καταλήξει ακόμα χειρότερα. Αν κοιτάξετε την όλη κατάσταση, είχαμε τρεις συναντήσεις μέχρι τον Οκτώβριο και άλλη μία τέταρτη τον Νοέμβριο και σε αυτές τις τέσσερις συνεδριάσεις συζητήθηκαν όλα τα σημεία τα οποία τελικά συμφωνήθηκαν στην Κοπενχάγη. Τώρα αν με ρωτάτε αν μπορούσαμε να είχαμε κάνει τα πράγματα διαφορετικά, ναι, ίσως ναι, αλλά δεν νομίζω ότι τελικά θα είχαμε επιτύχει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Γιατί ναι, πράγματι μπορείτε να επιλέξετε το ένα ή το άλλο πράγμα και να πείτε ότι εάν το είχαμε κάνει αλλιώς, ίσως να. Αλλά όλοι όσοι ήταν εκεί συμφωνούν ότι ανεξάρτητα από το τι είχαμε τελικά κάνει, κάποιες χώρες άλλαξαν την στρατηγική τους και στο τέλος της όλης διαδικασίας αποφάσισαν ότι δεν επιθυμούν συμφωνία. Δεν μπορώ να μπω στις λεπτομέρειες γιατί δεν έχω χρόνο στη διάθεσή μου, αλλά αυτή είναι η άποψή μου για το θέμα. Εάν δεν είχαμε αυτήν την στεναρή θέση, τότε οι άλλες χώρες μπορεί να είχαν τελικά πολύ διαφορετική προσέγγιση. Και θα ήθελα, θα ήθελα αν βρείτε μια οποιαδήποτε άλλη προεδρία προηγούμενη που να είχε βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες, να είχε κάνει περισσότερες ε, επισκέψεις, αν υπήρχε άλλη προσπάθεια για να συνεργαστούν, θα σας δώσω μια σαμπάνια. Δεύτερο ερώτημα. Δεν είμαστε εδώ ε, για αυτό το σκοπό, αλλά για να συνεργαστούμε. Μπορείτε όμως να μας πείτε ένα σφάλμα, όχι τρία, ένα. Όχι μόνο στην ε, Δανική Προεδρία, αλλά γενικότερα στην Ένωση. Εδώ μιλάμε για τη δύσκολη θέση στην οποία βρισκόμαστε, γιατί δεν μιλάμε με μία φωνή. Και τι θα κάνετε για να το νικήσετε αυτό, πώς θα, θα φημώσετε τον κύριο Σαρκοζή, τι, τι προτίθεστε να κάνετε όταν όλοι κάνουν δηλώσεις σε διεθνές επίπεδο για τα θέματα κλίματος. Απάντηση. Για αυτό το τελευταίο δεν νομίζω. Τώρα, δεν νομίζω ότι πρόβλημα της Ένωσης είναι ότι μιλάει με διαφορετικές αλλά είναι όταν είμαστε σε μία αίθουσα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, με τον Κινέζο. Εκεί είναι το πρόβλημα. Το ότι είναι πολλοί όσοι εκπροσωπούνται στη, από την Ευρώπη δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Καλύτερο είναι να μιλάνε με μία φωνή. Αλλά νομίζω ότι... Δεν νομίζω ότι κάποιος θα είχε πετύχει καλύτερα αποτέλεσμα από αυτό ανεξάρτητα από το ποιος θα ήταν αυτός που θα εξέφραζε αυτήν την νέα φωνή, σοβαρά πρέπει να σκεφτούμε ποια είναι πραγματικά η θέση μας στον κόσμο. Νομίζω ότι κανένας δεν θα ακούσει το τι λέει η Ευρώπη εάν δεν μιλάμε με μία φωνή για τόσο ζωτικής φύσεως θέματα. <laughs> Το να εμποδίσει κανείς τον Σαρκοζή να λέει αυτά που λέει, αυτό είναι κάτι το ανέφικτο, το αδύνατο μάλλον. Ο κ. Σκυλακάκης έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ. Ε, Πρόεδρε, κύριε υποψήφιε επίτροπη, για το mainstreaming μπορείτε να διευκρινίσετε αν θα ε, εισάγετε αξιολόγηση των επιπτώσεων στη μελλοντική κλιματική νομοθεσία. Στην αναθεώρηση του κοινοτικού προϋπολογισμού θα ε, έχετε μια διαδικασία ελέγχου. Θα ξεκινήσετε έναν διαγνωστικό έλεγχο της σημερινής πολιτικής ε, και θα μας δώσετε και κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα για όλα αυτά. Θα πρέπει να υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές για, την, για τους κανόνες προμήθειας για κλιματικά θέματα. Θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στη δασική πολιτική, γιατί χάνουμε ε, και θα χάσουμε τις επόμενα, τα επόμενα 20-30 χρόνια ε, δισεκατομμύρια εκτάρια και οι κρατικές επιδοτήσεις για τον άνθρακα θα αναθεωρηθούν την κλιματική αλλαγή, θα την εντάξετε σε αυτή την πολιτική. Σε μία ερώτηση α, δεν μπορώ να απαντήσω σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Η μελέτη αντικτύπου είναι πολύ σημαντική, ίσως όχι σε όλα, γιατί θα πρέπει να προσέξουμε να μην κάνουμε τέτοιες μελέτες όταν δεν χρειάζονται. Αλλά ανέφερα ήδη στην αρχή ότι ο κλιματικός έλεγχος, μια και η Ένωση πληρώνει με τα διάφορα ταμεία, ε, είναι λογικό να προσέξουμε ότι όταν υπάρχει κοινοτική χρηματοδότηση θα πρέπει να, ελέγχουμε ότι ξοδεύουμε τα χρήματα ανάλογα. Θα πρέπει να έχουμε έναν οδικό χάρτη για τις επόμενες δεκαετίες και αν δεν υπάρχει αυτό ο έλεγχος στην αρχή, τελικά ξοδεύουμε εκ των υστέρων πάρα πολλά λεφτά από του φορολογούμενους. Ε, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να διορθωθεί λοιπόν. Επίση, θα πρέπει να έχουμε ένα κλιματικό και μεταφορικό πακέτο ε, μαζί με τον Επίτροπο Μεταφορών για να δούμε σε ποιου τομεί μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε. Ε, ε για τι εκπομπέ των αυτοκινήτων, διαγνωστικό έλεγχο ναι, επίσης οι προμήθειες θα πρέπει να, έχουν, να γίνουν πιο πράσινες. Υπάρχουν τόσοι τομείς όπου οι διάφοροι δημόσιοι τομείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαν να είχαν βοηθήσει για να κινηθεί προς σωστή κατεύθυνση η αγορά. Δεν χρησιμοποιούμε αυτές τις δυνατότητες σωστά. Η δασική στρατηγική είναι πολύ σημαντικό, θα το συζητήσω με τον κύριο Ποτότσνικ. Ε, Πραγματικά είναι προβληματικό που δεν καταφέραμε να έχουμε ευρωπαϊκή θέση για ως Ευρώπη μέχρι την COP15. Νομίζω ότι είναι ένας τομέας που πραγματικά υπάρχει καθυστέρηση. Θα επανέλθω στη μόνη ερώτηση που δεν απαντήσατε. Μπράβο που απαντήσατε στις υπόλοιπες. Ε, στις ε, επιδοτήσεις ε, για τα καύσιμα. Ξοδεύουμε παγκόσμια 300 ε, δισεκατομμύρια για να επιδοτήσουμε, να επιχορηγήσουμε τα ορυκτά καύσιμα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και δεν έχουμε πολιτική, πραγματική πολιτική γι' αυτό. Γιατί και εμείς το ίδιο κάνουμε και εμείς επιδοτούμε. Αυτό είναι θέμα της εντολής σας. Δεν νομίζω ότι πρέπει να επιδοτούμε τα καύσιμα. Ήταν και τμήμα της δήλωσης του G8, αν θυμάμαι καλά φέτος το καλοκαίρι στην, στο Άκυλα. Είπαμε ότι παγκόσμια δεν πρέπει να επιδοτούμε τα καύσιμα. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να το κάνουμε αυτό. Ε, γιατί πολλές αναπτυσσόμενες χώρες κινούνται προς άλλη κατεύθυνση και θα χρειαστεί χρόνος. Αλλά αν θέλουμε να είμαστε λιγότερο εξαρτημένοι από τα ρηκτά καύσιμα, όλοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν είναι σόφρον να επιδοτούμε αυτά τα καύσιμα. Ευχαριστώ πολύ. Ερχόμαστε στο πρώτο ερώτημα από την Επιτροπή Βιομηχανίας. Ε, έχουμε έχει, ο συνάδελφος έχει συνοψίσει έξι ερωτήσεις σε μία. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ καλό γιατί επιτρέπει στην Επιτροπή Βιομηχανίας να παρουσιάσει όλα αυτά τα ερωτήματα από κοινού. Έχουμε τον κύριο Μπένσεν, λοιπόν, ο οποίος θα λάβει το λόγο. Καλώς ήλθατε στις Βρυξέλλες καταρχήν. Νομίζω ότι έχετε κάνει εξαίρετη εργασία ως, επιτροπός, ως Υπουργός μάλλον, Περιβάλλοντος της Δανίας και στη συνέχεια σαν Υπουργός Κλίματος και Ενεργείας. Είναι λυπηρό βέβαια για όλους μας ότι δεν καταφέραμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία μεταξύ των COP15 για την Κοπενχάγη. Και το αποτέλεσμα της Κοπενχάγης δεν σημαίνει ότι σταματάει ο κόσμος να γυρίζει, απλώς ότι πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπαθίες μας για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Η Ευρώπη θα πρέπει να αναπτύξει πράσινες τεχνολογίες, βιώσιμες τεχνολογίες, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και νέες θέσεις που να είναι πράσινες. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να ανταγωνιστούμε <clears throat> τα ημερομίσθια άλλων χωρών. Εγώ φοβάμαι ότι έχουμε ένα πρόβλημα δημιουργία θέσεων απασχόληση. Τι θα κάνετε για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε αυτή την ε, πρόκληση που σημαίνει να κάνουμε κάποιες πρόοδους για την έρευνα και την τεχνολογία στις πράσινες ενέργειες. Η απάντηση. Εγώ θα ήθελα <clears throat> να δώσω ιδιαίτερη έμφαση στην ε, έρευνα είναι ένα πρόβλημα το ότι είμαστε 27 χώρες και όχι μία χώρα μονάχα που εργάζεται στο θέμα αυτό. Είναι απαραίτητο λοιπόν να μπορούμε να έχουμε ένα πιο συστηματικό τρόπο αντιμετώπιση, ιδίω όταν πρόκειται για οικονομική αναδιάθρωση. Συγχρόνω όμω θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα δυνατά σημεία τα οποία έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία μπορούμε να προωθήσουμε με κοινή έρευνα. Περισσότερα προγράμματα επίδειξη, παραδείγματο χάρη. Αυτό είναι μια τεράστια πρόκληση. Να περάσουμε από τη φάση που έχει κανεί απλώ μια καλή ιδέα σε ένα κέντρο έρευνα μέχρι ότου αυτό γίνεται κάτι το οποίο μπορεί να περάσει στην φάση εμπορία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μαύρη τρύπα μεταξύ της έρευνας και της εφαρμογής. Και υπάρχει και το πρόβλημα της χρηματοδότησης ώστε η Ευρώπη να μπορεί να προωθεί αυτά τα προϊόντα. Είναι ακόμα πολύ χαμηλός ο προϋπολογισμός έρευνας στην Ευρώπη. Κάτι ακόμα το οποίο είναι σημαντικό είναι το πώς μπορούμε να αποφύγουμε να επικεντρώνουμε πάντα την προσοχή μας στις μεγάλες επιχειρήσεις, στους μεγάλους παίκτες στην ευρωπαϊκή οικονομία. Γιατί η ευρωπαϊκή οικονομία στο μεγαλύτερο μέρος της αποτελείται από μικρομεσαίες εταιρείε και επιχειρήσεις. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σε επαφή με τους εκπροσώπους τους για να δούμε πώς μπορεί να κάνει τι μπορεί να κάνουν μικρές εταιρείε για να λύσουν προβλήματα του περιβάλλοντος. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να εμπνευστεί από θετικές πρακτικές οι οποίες μπορούν στη συνέχεια να, α, να εφαρμοστούν με τη βοήθεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τόμψον. Ευχαριστώ. Και εγώ σας καλωσορίζω στις Βρυξέλλες. Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα της πυρηνικής ενέργειας. Γιατί όταν συζητήσαμε την οδηγία, συζητούσαμε την οδηγία για τους δεσμευτικούς 2020, 2020-2020. πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πολλοί υπουργοί ζήτησαν η πράσινη ενέργεια και η πυρηνική ενέργεια να προωθηθούν γιατί έχουν μικρότερες ε, εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Όταν οι υποψήφοι επίτροποι έρευνας και ενέργειας ήρθαν εδώ, είπαν και οι δύο ότι η πυρηνική ενέργεια είναι πολύ σημαντικό τρόπο για να μειώσουμε τι εκπομπέ του διοξείδου του άνθρακα και αν θα συνεχιστεί η έρευνα προ αυτή την κατεύθυνση. Εσεί όμω ε, είπατε ότι έχετε κάπω αποστασιοποιηθεί από την πυρηνική ενέργεια. Ε, θα θέσετε βέτο λοιπόν για την πυρηνική ενέργεια ε, και σε αυτό το επιχείρημα ότι μειώνει τι εκπομπέ του διοξείδου του άνθρακα. Και θα θέσετε βέτο για την έρευνα για την πυρηνική ενέργεια. Όχι. Όχι, όχι, λέει η υποψήφια επίτροπο. Αυτό που εννοούσα είναι ότι δεν αποστασιοποιήθηκα στην πραγματικότητα από την πυρηνική ενέργεια. Στη Δανία, στη χώρα μου, λάβαμε εκεί κάποιε αποφάσει και είπαμε ότι δεν θέλουμε πυρηνική ενέργεια. Κάναμε μια άλλη ουσιαστική ε, επιλογή. Και νομίζω ότι το είπα και στην πρώτη μου απάντηση ότι η πυρηνική ενέργεια, η πυρηνική ενέργεια υπάρχει στον κόσμο. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει ασφάλεια και ότι υπάρχουν νέες γενιές ε, αντιδραστήρων. Και το πρόβλημα των πυρηνικών αποβλήτων ε, μειώνεται λόγω των νέων αυτών γενιών ε, αντιδραστήρων. Για τα θέματα της δικής μου αρμοδιότητας θέλω να πω ότι η πυρηνική ενέργεια υπάρχει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει έρευνα σε αυτόν τον τομέα. Θα είμαι πολύ προσεκτική όμως χρησιμοποιούμε πάρα πολλά χρήματα για αυτή την έρευνα και πολύ λιγότερα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό είναι που δεν μου αρέσει. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μην επενδύουμε υπερβολικά και δυσανάλογα στην πυρηνική ενέργεια και λιγότερο στις υπόλοιπες μορφές ενέργειας. Νομίζω ότι θα πρέπει να κατανείμουμε διαφορετικά τα χρήματα. Είναι πολύ σημαντικό σε ένα τομέα ότι στον τομέα των ε, ανανεώσιμων, πηγών ενέργειας θα πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερες προσπάθειες. Ο Ιβο Μπέλετ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία <clears throat> Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υποψήφια Επίτροπε, εδώ είμαι. Θα σας θέσω ένα ερώτημα στα Ολλανδικά για τα υπεράκτια σχέδια ε, δικτύων ενεργείας στη Βόρεια Θάλασσα υπάρχει αυτό το γιγάντιο σχέδιο το οποίο έχει ξεκινήσει η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο και άλλες έξι χώρες ουσιαστικά θα συμμετάσχουν, θα κοστίσει δεκάδες δισεκατομμυρίων ευρώ. Ένα συγκεκριμένο ερώτημα για αυτά τα ενεργειακά δίκτυα. Φαντάζομαι ότι τα υποστηρίζετε κι εσείς. Πώς συγκεκριμένα θα υποστηρίξετε τα προγράμματα αυτά ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρησιμοποιήσετε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία θα προτείνετε και τα οποία θα, θα, θα διεκδικήσετε χρηματοδότηση για αυτά έναντι των συναδέλφων σας και ποια είναι η άποψή σας για την ιδέα του να επιτρέψουμε σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες να έχουν την δυνατότητα χρηματοδοτικά να συμμετάσχουν σε αυτά τα σχέδια και να μπορέσουν να αποκομίσουν μερίσματα από αυτά. Νομίζω ότι αυτό το δίκτυο ενέργειας είναι ένα από τα πιο αποδοτικά που μπορούμε να δημιουργήσουμε. Όσο πιο αποδοτικά είναι τα δίκτυα, τόσο και καλύτερα. Αν μπορούμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε μεγάλη απόδοση ενέργειας, εγώ είχα συμμετάσχει λίγο ως υπουργό Ενέργειας στο, στην προετοιμασία αυτού του σχεδίου, το οποίο δίνει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία στα ενεργειακά μας συστήματα. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε λοιπόν αυτή την ευελιξία μέσω της χρήσης ενός μεγαλύτερου ποσοστού ανανεώσιμης ενέργειας. Εγώ δεν ξέρω τις λεπτομέρειες για αυτά τα σχέδια. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι στο χαρτοφυλάκιο του Επιτρόπου Ενέργειας. Εγώ δεν εμπλέκομαι άμεσα για αυτό το θέμα και επομένως δεν μπορώ να σας δώσω μια πλήρη και μακροσκελή απάντηση. Ευχαριστώ. Τρίτος γύρος ερωτήσεων. Η κυρία Χίμπνερ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε, κυρία υποψήφια επίτροπε. στην πρόσφατη διάσκεψη κορυφής στην Κοπενχάγη παρά τις προσπάθειες της Ένωσης για επιτυχία δεν υπογράφηκε καμία συγκεκριμένη δέσμευση για παγκόσμια μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου. Και κυρίως εξαιτία της θέσης της Κίνας και της Ινδίας. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει στις διεθνείς διαπραγματεύσεις να έχει την ίδια πολιτική γραμμή ή να είναι πιο ευέλικτη εναντί των χωρών αυτών. Και δεύτερον, τι πιστεύετε για αυτήν την κλοπή των mail από το ερευνητικό κέντρο. Απάντηση. Σε ό,τι αφορά το Climate Gate, ξέρω ότι ο πρόεδρος κ. Πιτουρή στην Κοπενχάγη υποσχέθηκε να εξετάσει το θέμα, αλλά εγώ πιστεύω ότι για μένα δεν αλλάζει τίποτα. Κατά καιρού μπορούν να διαρρεύσουν διάφορα mail. Αλλά μιλάμε εδώ για πολλούς χιλιάδες ερευνητές που γνωρίζουν πολύ καλά τι συμβαίνει και μας συμβουλεύουν. Και δεν νομίζω ότι όλα αυτά θα αλλάξουν μόνο και μόνο επειδή διαρρέει κάποιο είδους ανταπόκριση με mail. Επίσης πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να είμαστε και πολύ αρνητικοί για τα όσα συνέβησαν με τις μεγάλες οικονομίες στην Κοπενχάγη. Και μάλιστα εγώ τα βλέπω αλλιώς. Η Βραζιλία μερικέ εβδομάδε πριν την Κοπεχάγη έθεσαν εθνικό στόχο και παρά τα αποτελέσματα της Κοπενχάγης θα προσπαθήσουν να μειώσουν τις εκπομπές τους κατά 35 έως 38%. Αυτό είναι πολύ ουσιαστικό για μια οικονομία όπως τη Βραζιλία. Και η Κίνα είπε ότι θα μειώσει κατά 40 με 45% θα ήθελα και ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, αλλά για, μια, για τόσο μεγάλες οικονομίες και να παρεκκλίνουν των πενταετών προγραμμάτων και να πούν ότι μέχρι το 2015-2020 αυτό θα κάνουμε, μας δείχνει αυτό ότι είναι σοβαροί στις προσπάθειές τους. Δηλαδή, ναι, έχετε δίκιο, δεν υπογράφηκαν δεσμεύσεις, αλλά στην συμφωνία της Κοπενχάγης λέει ότι θα καταστήσουν, θα κάνουν ενεργειακές δράσεις και θα ελεγχθεί ό,τι έχουν αποτελέσματα στη χώρα τους. Είναι λοιπόν ένα σημαντικό πρώτο βήμα. Στο Κιώτο η ΙΠΑ, η Βραζιλία, η Κίνα, η, Ινδία δεν ήταν μέλος οποιασδήποτε υποχρέωση. Τώρα όμως λένε ότι για να επιλύσουμε παγκοσμίω το πρόβλημα πρέπει να έχουμε παγκόσμια ευθύνη. Μία ένα σύντομο συμπληρωματικό ερώτημα, κάτι το οποίο ήδη θίξατε. Προβλέπετε μία συνάντηση για να διερευνηθεί το όλο θέμα των ε, mail που έχουν γίνει αντικείμενο διαρροής και να ελεγχθεί το περιεχόμενό τους. Απάντηση. Οι ίδιοι επιστήμονες θα πρέπει να ασχοληθούν με αυτό. Στην ουσία εμείς ως πολιτικοί έχουμε μόνο μία επιλογή. Μπορούμε να αποφασίσουμε. Θέλουμε να ακούσουμε την επιστήμη η οποία μας λέει ότι εάν διστάσουμε διατρέχουμε τεράστιο κίνδυνο εις βάρος των μελλοντικών γενεών. Αυτό είναι το ένα. Ή μπορούμε να πούμε εντάξει. Σε 20-30 χρόνια οι επιστήμονες θα μας πούν σε κάτι διαφορετικό. Τι θα ήταν χειρότερο. Να είχαμε επιτύχει τελικά πιο αποτελεσματικές κατά, καθαρές τεχνολογίες, να είμαστε λιγότερο εξαρτημένοι από τα καύσια. Δηλαδή ακόμα και αν δεν το πιστεύετε και είστε σκεπτικιστής για τις κλιματικές αλλαγές, μήπως όλα αυτά τελικά θα είναι καλύτερες ιδέες όταν θα έχουμε γίνει 9 δισεκατομμύριο και θα έχουμε μειωμένους σπόρους. Euh, Ο κύριος Παρνιό. Ε, Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, προηγουμένως είπαμε ότι μετά την αποτυχία της διάσκεψης στην Κοπενχάγη, η κοινή γνώμη στην Ευρώπη κατέστη αυστηρή. Θεωρεί ότι η Κοπενχάγη είναι και αποτυχία και επίσης πιστεύει ότι αυτοί που θα πρέπει να πληρώσουν πιο ακριβά το τίμημα τελικά είναι αυτοί που είναι τα μεγαλύτερα θύματα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Πρέπει να αποκατασταθεί μια εμπιστοσύνη εν ώψη της ε, διάσκεψης του Μεξικού. Θα πρέπει ε, να, να ανακτήσουμε αυτή την, ε, την ηγεσία, τον ηγετικό ρόλο ως Ευρώπη, προτείνοντας όμως θεσμευτικά οικονομικά μέτρα. Για πρώτη φορά λοιπόν σήμερα το πρωί έχετε την ευκαιρία εν ονόματι της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παίξετε αυτό τον ηγετικό ρόλο και να μας πείτε ποια είναι η δική σας πρόταση, ούτω ώστε να υπάρξει αυτή η εμπιστοσύνη, να αποκατασταθεί αυτή η εμπιστοσύνη, ε, προτείνοντας, Φερρυπίν, όπως κάποιοι, ε, ένα φόρο στα σύνορα της Ευρώπης ή ένα πράσινο φόρο, όπως προτείνουν άλλοι, για τα προϊόντα που προέρχονται από χώρες που δεν σέβονται τους περιβαλλοντικούς κανόνες. Ή μια άλλη πρόταση που υπάρχει, ένα φόρο για το διοξίδιο του άνθρακα, ε, στις συναλλαγές. Πέστε μας, εσείς, τι πρόταση έχετε να κάνετε. Ποια είναι η θέση σας. Καταλαβαίνω την ανησυχία σας. Ε, η κοινή γνώμη έχει αφυπνιστεί. Δεν έχουμε φτάσει στους στόχους μας, ε, πώς μπορούμε να κρατήσουμε αφυπνισμένη αυτή την κοινή γνώμη και πώς θα εξασφαλίσουμε δεν θα πληρώσουμε μόνοι το τίμημα. Ε, Επίση, έχετε δίκιο να μιλάτε για την οικονομική κρίση και τι επιπτώσει τη. Αλλά αν ε, με συνετό τρόπο βγούμε από την οικονομική κρίση, μπορούμε να ε, καλύψουμε ε, επενδύοντας κάποιες από τις θέσεις απασχόλησης που χάσαμε. Για να δείξουμε στον κόσμο ότι η ατζέντα μας δεν είναι εναντίον των θέσεων απασχόλησης. Το θέμα είναι να έχουμε μια πιο έξυπνη ανάπτυξη. Ξέρω την συζήτηση για το φόρο για το διοξίδιο του άνθρακα. Σε ορισμένε χώρες θα υπάρχει τέτοιο φόρος για τους τομείς που δεν καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Αλλά εγώ πιστεύω ότι τώρα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε ούτως ώστε να περάσει αυτή, να υπάρξει αυτή η διεθνή συμφωνία που θα είναι η πρώτη μας προτεραιότητα για το Μεξικό, μέχρι να φτάσουμε στο Μεξικό. Και μετά να φτάσουμε στον ελάχιστο κοινό παρανομαστή, παραδείγματος χάρη αυτό το τέλος στα σύνορα, το φόρο στα σύνορα. Παραδείγματο χάρη, το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών δέχεται το σύστημα. Η Ιαπωνία θα κάνει το ίδιο του χρόνου. Η Αυστραλία η Νέα Ζηλανδία είπε ότι θα έχουν ένα σύστημα εμπορίας εκπομπών. Νομίζω ότι αυτό είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος. Και η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία προτιμάει αυτή τη λύση παρά τις άλλες λύσεις, γιατί είναι και περιβαλλοντικά αποτελεσματική και δίνει και τα σωστά κίνητρα για να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Θα ήταν λάθο ε, χρονική στιγμή να πούμε τώρα ότι πάμε στου φόρου και στα τέλη. Αργότερα θα μπορούσαμε να καταφύγουμε εκεί, αν δεν καταφέρουμε αυτό που μας ενδιαφέρει πιο πολύ, την ε, Διεθνή Συμφωνία. Η διαρροή του άνθρακα σίγουρα ε, ενδιαφέρει πάρα πολύ τις ευρωπαϊκές αγορές και τις θέσεις απασχόλησης. Ε, πέρα από τη βιομηχανία όμως, τις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα πρέπει κάπως να καθησυχάσουμε και τους εργαζόμενους, οι οποίοι ανησυχούν τα μάλα. Δεν σας κατάλαβα από τη διερμηνία. Είπατε ότι η διαρροή του άνθρακα θα μας απασχολήσει σε ό,τι αφορά την, τις θέσεις απασχόλησης. Ε, την εμπιστοσύνη αυτή μπορούμε να τη δώσουμε στους εργαζομένους που μετά την Κοπενχάγη θεωρούν ότι υπάρχει αδικία. Θα πρέπει να τους δώσουμε κάποιες προοπτικές, ούτως ώστε να τους επιτρέψουμε να πούν ότι τα έσοδα που αποκομίζουμε από αυτές τις πολιτικές ε, δεν είναι εις βάρος τους και τα ωφέλη που αποκομίζουμε από αυτές τις πολιτικές. Καταλαβαίνω αυτή την ανησυχία για τη διαρροή του άνθρακα και τις μετεγκαταστάσεις δηλαδή. Αλλά πιστεύω ότι αν φοβηθούμε τώρα αυτή είναι συνταγή αποτυχίας. Γιατί πραγματικά θα υπάρχει, θα υπάρχει πρόβλημα με τις θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος. Και να σας πω γιατί μπορούμε να δημιουργήσουμε τις απασχόλησεις με αυτές τις πολιτικές. Στη Δανία το 2008, την τελευταία εντό αγωγικών κανονική χρονιά πριν την κρίση, η ενεργειακή αποτελεσματικότητα και η εξαγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αυξήθηκε κατά 19%. Στη χώρα μου, ο κόσμος πείθεται εύκολα ότι αν τα καταφέρουμε, θα κερδίσουμε και θέσεις απασχόλησης. Θα υπάρξουν έσοδα από τις αυξημένες εξαγωγές. Το θέμα είναι να, να κάνουμε όλη αυτή την προσπάθεια σωστά. Σύπα είναι το θέτει το επόμενο ερώτημα. Σωστά είπατε ότι χρειαζόμαστε πράσινη ανάπτυξη και το ότι πρέπει να βοηθήσουμε την βιομηχανία μας να αλλάξει, να είναι ανταγωνιστική στο μέλλον. Δεν φοβάμαι εγώ στην ουσία την διαρροή άνθρακα, γιατί στην ουσία οι επιχειρήσεις δεν πάνε σε χώρες με χειρότερες υπηρεσίες και χειρότερη νομοθεσία, αλλά φοβάμαι ότι δεν τους βοηθάμε στην ουσία να αλλάξουν αποδοτικά και όσο γρήγορα απαιτείται. Και είπατε κι εσείς ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση. Πώς όμως, υπάρχει ίσως κίνδυνος ότι τώρα που έχουμε τη στρατηγική για το 2020 γίνονται πολλά λόγια. Πολλές φορές μιλάμε για την πράσινη ανάπτυξη, αλλά μας λείπουν τα εργαλεία. Και χρειάζεται πιο βιώσιμη και σωστή χρήση πόρων και ενέργειας. Ρωτώ λοιπόν πώς θα το εξασφαλίσετε αυτό και ποια είναι τα εργαλεία που θα χρησιμοποιείτε, κλιματικός έλεγχος, επιδόσεις κτλ. Πιστεύω ότι το σύστημα εμπορίας εκπομπών είναι πολύ αποτελεσματικό εργαλείο. Γιατί αν είστε μη αποτελεσματικός, πληρώνετε ένα πολύ ακριβό τίμημα. Υπάρχει λοιπόν μεγάλο κίνητρο για να ξανασκεφτείτε τον τρόπο παραγωγής σας, να βελτιώσετε το αύριο. Αυτό λοιπόν είναι και ένα όριο. Θα χθεσπίσουμε 50 διαφορετικά benchmarks που θα καλύπτουν μεγάλο τμήμα της βιομηχανίας και αυτό θα θεωρηθεί πλέον όχι ως βάρος αλλά και ως έμπνευση. Πώς μπορούμε να αντιγράψουμε τους καλύτερους από μας. Και επίσης πιστεύω ότι για τις επιχειρήσεις και την βιομηχανία πρέπει να είμαστε πολύ πιο εστιασμένοι ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την έρευνα και τα προγράμματα επίδειξης. Μπορούμε επίσης να κάνουμε προσπάθειες και στον τομέα της εκπαίδευσης. Πριν μερικά χρόνια η Ευρώπη, στην Ευρώπη λέγανε ότι εμείς σχεδιάζουμε αυτά τα νέα προϊόντα και η Κίνα θα τα κατασκευάζει. Δεν νομίζω ότι έτσι είναι τα πράγματα ούτε καν σήμερα και είμαι σίγουρο ότι δεν θα είναι και έτσι αύριο. Νομίζω ότι θα πρέπει να επενδύσουμε πολύ στην επιχειρηματική δραστηριότητα, να δώσουμε κίνητρα σε αυτούς που επιχειρούν και η παιδεία μας και η εκπαίδευσή μας να βελτιωθεί. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και νομίζω ότι τελικά δεν είμαστε πολύ καλοί στην Ευρώπη να μοιραζόμαστε τις βέλτιστες πρακτικές. Στην Δανία είπαν κάποιοι Κάποιε βιομηχανίε ότι δεν μπορούν να συζητήσουν μεταξύ του γιατί είναι ανταγωνιστριε. Όμω, τώρα κατάλαβαν ότι είναι λογικό να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, να μάθουν η μία από την άλλη επιχείρηση και να είναι πιο ισχυρέ μετά για τι εξαγωγέ του. Νομίζω ότι μπορούμε να υποφεληθούμε από τα βέλτιστα παραδείγματα και τις ανταλλαγέ βέλτιστων πρακτικών. Ένα συμπληρωματικό ερώτημα. Πιο συγκεκριμένα, είστε διατεθειμένοι να προωθήσετε το eco-design για όλα τα προϊόντα και πώς θα προσμετρηθεί λογιστικά η παραγωγή άνθρακα των, επιχειρήσεων. Απάντηση. Η οδηγία για το eco-design είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν έχει δουλέψει τόσο γρήγορα όσο αναμείναμε ως δανείδη υπουργό. Κάθε έξι μήνες το κοιτούσα και κοιτούσα την πρόοδο, αλλά τελικά είναι αργή η πρόοδος αλλά θεωρώ ότι είναι αποτελεσματική. Θα εξετάσουμε το αν θα πρέπει να διευρυνθεί και δεν είμαι απόλυτα σίγουρη για το ποιε πρέπει να είναι, πρέπει να είναι οι περιορισμοί αλλά είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο και νομίζω ότι πρέπει να θέσουμε πρότυπα, να συνεργαστούμε. Το να θέσουμε πρότυπα είναι πολύ καλό εργαλείο στην Ευρώπη. Κοιτάξτε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Θα υπάρχει ανταγωνισμός αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αν προσπαθούμε να συντονιστούμε και να έχουμε τελικά πρότυπα τα οποία να είναι κοινά στο τέλος παρά να προσπαθούμε να καινοτομούμε ο ένας ενάντια στον άλλον. Ευχαριστώ. Ακολουθεί το πρώτο ερώτημα από την Επιτροπή Μεταφορών, ο κύριος Ιτελέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το ερώτημά μου αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές. Όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται για τις μεταφορές πρέπει να ληφθούν έχοντας ως γνώμονα και το περιβάλλον. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός έχει αποφασίσει να μειωθούν οι εκπομπές θείου, μάλλον το ποσοστό θείου στη, στα καύσιμα από 0,5% σε 0,1%. Αυτό αφορά μονάχα τη Βαλτική και τη Βόρεια Θάλασσα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια στρέβλωση ανταγωνισμού μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο δεν είναι απόλυτα δίκαιο. Με ποιο τρόπο που θα μπορούσαμε εμείς να συνδυάσουμε αυτές τις δύο πολιτικές, την πολιτική μεταφορών και την πολιτική περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα έπρεπε ίσω να αναβληθεί μια λήψη απόφαση για τα θέματα αυτά. Πώ θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα αντιμαχόμενα θέματα. Αν αυτό είναι μια ε, απόφαση του διεθνού Ναυτιλιακού Οργανισμού, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αν οι εμπλεκόμενε πλευρέ στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό το συμφώνησαν, θα πρέπει να το αποδεχτούμε και θα πρέπει να προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να εξασφαλίσουμε ότι η ρύθμιση του ναυτιλιακού τομέα γίνεται σε διεθνέ επίπεδο από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό ορισμένε φορέ έχει καθυστερήσει ο ναυτιλιακό οργανισμό στη λήψη αποφάσεων. Εγώ έχω συνεργαστεί μαζί του στο παρελθόν και η ελπίδα μου ήταν στην Κοπεχάγη να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που περιλαμβάνει τα θέματα τη διεθνού ναυτιλία και της των αεροπορικών μεταφορών. Και πρέπει να πω σαφέστατα προ την κατεύθυνση του Διεθνού Ναυτιλιακού Οργανισμού ότι ναι, με προτιμώ τι διεθνεί ρυθμίσεις, να αποφασίζονται σε διεθνές επίπεδο οι κανονιστικές ρυθμίσεις για την αυτιλία, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προχωρούν με ταχύτητα και όχι να συνεχίσουν να χρονοτριβούν και να διστάζουν. Και αυτό ισχύει και για την αυτιλία και εκεί ορισμένε φορές πρέπει να πιέσετε ένα τομέα για να εξυγχρονιστεί. Νομίζω ότι αυτό λειτουργεί και ξέρω ότι σε καιρό κρίσης πολλές από τις εταιρείες τις ναυτιλιακές αποφασίσει να κινηθούν οι ίδιες γιατί βλέπουν ότι είναι απόλυτα λογικό όχι μόνο για το περιβάλλον αλλά και οικονομικά. Ευχαριστώ. Ένα συμπληρωματικό ερώτημα. Στην περίπτωση της Βαλτικής, οι Ρώσοι οι οποίοι δεν συμμετέχουν, δεν θα εφαρμόσουν την απόφαση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού θα έχουν ένα πλεονέκτημα και θα κυριαρχήσουν στις ναυτικές μεταφορές στη Βαλτική. Επομένως, ουσιαστικά βάζουμε ένα αυτογκόλ. Ποια είναι η άποψή σα για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της Ρωσίας. <clears throat> Συμφωνώ μαζί σας ότι αυτό ισχύει πάντα για οποιαδήποτε ρύθμιση περιβάλλοντος που κάνουμε στη Βαλτική θάλασσα. Εγώ όμως έχω δει να υπάρχουν κάποιες τροποποίησεις στις θέσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Αν περιλαμβάνει και αυτό το συγκεκριμένο θέμα δεν το γνωρίζω. Αλλά έχω δει τους τελευταίους μήνες ότι ο πρόεδρος Μετβεντεφ αρχίζει να υιοθετεί και αυτό στην ατζέντα του περιβάλλοντος με πιο έντονο τρόπο από ό,τι στο παρελθόν είδαμε από τη Ρωσική Ομοσπονδία και ίσως αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το εξετάσουμε και μέσα στα πλαίσια του διαλόγου Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας και ίσως μπορούν να προέλθουν και κάποια αποτελέσματα από αυτή τη δράση. Ευχαριστώ πολύ. Τέταρτος γύρος ερωτήσεων και ξεκινούμε με την Κρίστα Κλάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Χέντεγκάρτ. <clears throat> Εδώ είπα, από την άλλη μεριά. η συνδιάσκεψη Κοφεχάγης δεν απέδωσε τους καρπούς τους οποίους προσδοκούσαμε. Εμείς είχαμε θέσει φιλόδοξους στόχους στην Ευρώπη και αυτό περιλάμβανε ακόμα και την ε, οδηγία για την εμπορία των εκπομπών. Εκεί αναφέρεται ότι θα πρέπει αυτή η οδηγία να προσαρμοστεί στις διεθνείς συμφωνίες. Βλέπετε τώρα την ανάγκη να υπάρξει αυτή η προσαρμογή στην οδηγία και ποια είναι τα συμπεράσματα τα οποία αντλείται σε σχέση με την συμφωνία που επήλθε για αυτή την οδηγία μετά από την κατάρρευση της Κομπεχάης. Θα προβείτε σε μια προτροποποίηση της ε, οδηγίας βάσει του άρθρου 10β ή του άρθρου 28. Είναι κάτι το απαραίτητο. Υπάρχουν και άλλοι οποίοι αναφέρθηκαν στα benchmark. Αν θεσπίσουμε benchmarks τα οποία βασίζονται στην ε, μέση απόδοση των δελτίστων, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει και η δυνατότητα οι καλύτερε αυτέ επιχειρήσει να παίρνουν τα πιστοποιητικά εκπομπών χωρί κανένα κόστο. Θα ισχύσει αυτό. Δεν νομίζω ότι μετά από την έλλειψη συμφωνία στην Κοπενχάγη εμεί θα πρέπει να αλλάξουμε την οδηγία. Αλλά το σύστημα εμπορία εκπομπών μα δίνει καλέ προοπτικέ για το μέλλον. Νομίζω ότι και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και κάποιοι υπουργοί τους τελευταίους μήνες, τον τελευταίο χρόνο γενικά, ήταν σε στενή επαφή με βουλευτές από το Αμερικάνικο Κογκρέσο και προσπάθησαν ε, να δουν πώς θα διαμορφωθεί το Αμερικανικό σύστημα. Υπάρχει λοιπόν ε, δυνατότητα το δικό μας σύστημα που ήταν επιτυχές να μεταφερθεί. Ε, έχει αναγνωριστεί ότι ήταν ε, πετυχημένο και μπορούμε να το συνδυάσουμε με το αμερικανικό σύστημα. Ε, μπορούμε να έχουμε λοιπόν μια παγκόσμια τιμή για τον ε, διοξείδιο του άνθρακα, για τα σημεία αναφοράς, για τα benchmark. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει επιστροφή κατά 100%. Όχι, οι εταιρείε θα πρέπει, θα πρέπει όντως ε, να κινηθούν και μόνες τους. Συμπληρωματικό ερώτημα. Εντάξει, μπορούμε να θεσπίσουμε τα benchmarks. Αλλά σε άλλους τομείς για τις εκπομπές ε, διοξείδου θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, είπατε, την γεωργία και την κτηνοτροφία. Αυτό θα περιπλέξει τα θέματα. Ξέρουμε ότι τα φυτά ε, απορροφούν διοξίδιο του άνθρακος και εκπέμπουν οξυγόνο, από την άλλη μεριά πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτή την οδηγία. Τι θα προκύψει τότε για την παραγωγή των ε, τροφίμων στη δική μας, στην περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν από μια τέτοια συμπερίληψη. Είναι πολύ τεχνικό αυτό το ερώτημα για το πώς μετράμε το σημείο αυτό. Αλλά Υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι για να μετρήσουμε τις εκπομπές της γεωργίας. Στη Δανία, ας πούμε, έχουμε ένα σχέδιο για την πράσινη γεωργία, όπως λέμε. Ε, αν αλλάξουμε τον τρόπο παραγωγής, θα πρέπει να έχουμε κάποιους κανόνες για το πότε, ας πούμε, ε, θα έχουμε τις οδιές ε, το χειμώνα, ε, πώς θα βάζουμε τα φυτοφάρμακα με πιο αποτελεσματικό τρόπο, τέτοιου τύπου πράγματα. Φυσικά είναι πολύ δύσκολο, είναι μια ολόκληρη επιστήμη για να δούμε ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές ε, από κλιματική άποψης, αλλά υπάρχει δυνατότητα μέτρησης αν κρατήσουμε ας πούμε τις εκπομπές στο έδαφος. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε Διάφορε μεθόδους και θα πρέπει στο μέλλον να δούμε πώς ε, θα λειτουργήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν ε, δυνατότητες που μόνο, μέχρι στιγμής μόνο η Δανία και η Πορτογαλία έχουν χρησιμοποιήσει. Η Λίντα Μακάβεν τώρα. Κοιτάξτε προς τα αριστερά σας. Θα ήθελα και εγώ να μιλήσω για το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Στο εισαγωγικό σας σχόλιο μιλήσατε για τις μεταφορές και τις εκπομπές που αυξάνουν. Μιλήσατε και για την αυσιπλοεία. Στην οδηγία υπάρχει μια δέσμευση μέχρι το 2011 να υπάρξει κάτι και για την αυσιπλοεία, αν δεν υπάρξει διεθνή συμφωνία. Θα το, θα, νομίζω ότι θα πρέπει να το σεβαστούμε. Ε, για τις χερσαίες μεταφορές δεν υπάρχει στο σύστημα εμπορίας, ε, δεν υπάρχουν αυτές οι χερσαίες μεταφορές. Ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουμε ε, την ε, φορολόγηση στην πηγή. Στην Αυστραλία γίνεται μια μελέτη για τις χερσαίες μεταφορές. Τι άποψη έχετε. Καταρχάς θα πρέπει να σεβαστούμε το, την ημερομηνία του 2011 για την αυσιπλοεία. Όπως είπα και πριν, ε, θα πρέπει να πούμε ξεκάθαρα στη Διεθνή Ναυτιλιακή Οργάνωση ότι δεν έχουμε πια χρόνο. Αν μπορούν να κινηθούν λίγο πιο γρήγορα, κάνει ένα πρόβλημα. Δεν, δεν επιμένονται και καλά να τα ρυθμίσουμε αυτά τα πράγματα στην Ευρώπη. Ε, η ναυσιπλοεία είναι διεθνή τομέα ούτω ή άλλω. Και είναι πολύ εύκολα η βιομηχανία απλώ να πάρει μια άλλη. σημαία. Κάποια πλοία να πάρουν σημαίε ξένε, α πούμε. Καλό θα ήταν λοιπόν αν μπορούσε ε, ο Διεθνή Οργανισμό ε, Ναυτιλία να κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει, αλλά πρέπει λίγο να βιαστεί. Να κινηθεί με πιο γρήγορου ρυθμού. Τώρα, αν θα πρέπει να διευρύνουμε τη βάση του συστήματος εμπορίας εκπομπών. Η έκθεση Florence λέει ότι ίσως θα πρέπει να το κάνουμε. Ίσως θα πρέπει να έχουμε σκεφτεί τι σημαίνει αυτό για τη συμμετοχή των άλλων τομέων. Γιατί ο τρόπος που έχουμε διαμορφώσει το κλιματικό πακέτο αφήνει τα εθνικά αφήνει τα κράτη να προωθήσουν τις δικές σου εθνικές πολιτικές για τις μεταφορές. Διάφορες χώρες έχουν αρχίσει να έχουν ε, σύστημα να έχουν κάποιους τομείς οι οποίοι καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας εκπομπών και κάποιους τομείς όχι. Υπάρχουν εθνικά σχέδια λοιπόν ε, εγώ νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις μεταφορές, γιατί δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση των μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν συμπεριλάβουμε και τις μεταφορές στο σύστημα εμπορία εκπομπών και να, να το αντιμετωπίσουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο αυτό το θέμα. Όλοι πρέπει να κάνουν τις προσπάθειές τους ε, για να καταπολεμήσουμε τι κλιματικέ αλλαγέ. Θα σα κάνω την ερώτηση που έκανα ε, στον κύριο Ποτότσνικ. Εσεί τι θα αλλάζετε στον τρόπο ζωή σα για να συνεισφέρετε και εσεί σε αυτόν τον αγώνα. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Μου κάνανε αυτή την ερώτηση και ως ε, Υπουργό Κλίματος και ήταν πάντα δύσκολη ερώτηση. Και τώρα μου την κάνετε ως υποψήφια επίτροπο περιβάλλοντο: ε, ως ιδιώτης κάνω πράγματα που κάνουν και πολλές άλλες οικογένειες. Δεν είμαι ιστερική. Αλλά σιγά σιγά κάνω μικροπράγματα. Αγοράζω, ας πούμε, α, όταν αγόρασα καινούργιο αυτοκίνητο, α, αγόρασα ένα αυτοκίνητο της κατηγορίας Α, αντικαθιστώντας ε, το παλιό, παλιότατο αυτοκίνητο που είχα. Ε, επίσης, ε, βελτιώνω τη μόνωση του σπιτιού. Το Δεκέμβριο αντικαταστήσαμε κάποια παράθυρα με καινούρια, πιο αποτελεσμα... αποδοτικά ενεργειακά. Κοιτάζω την, τις ετικέτες και βλέπω και τα ενεργειακά θέματα. Ε, αυτά είναι πρακτικά ζητήματα που μπορεί να κάνει ο καθένας ας πούμε, στην καθημερινή του ζωή με μεγαλύτερη συνείδηση. Ωραία. Θα επανέλθει μάλλον αυτό το ερώτημα σε επόμενες ε, δύο ώρες. Ο Μπόγκος Λαυσόνικ έχει το λόγο. Εδώ είμαι. Ευχαριστώ. Η Ανατολική Ευρώπη <clears throat> παράγει πάνω από 90% της ενέργειάς της από τον άνθρακα. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτό θα οδηγούσε σε τεράστιο άχθος για τους πολίτες των χωρών αυτών και θα κατέστρεφε τις βιομηχανίες μας. Μπορείτε να λάβετε υπόψη το γεγονός ότι το κόστος της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να κατανεμηθεί εξίσου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ποιο τρόπο θα εξασφαλίσετε ότι θα υπάρξει ισοδίκαιος τρόπος κατανομής του κόστους και τι έχετε να πείτε για την ε, ενέργεια από καθαρή καύση άνθρακος. Πότε μπορούν να εισαχθούν σε βιομηχανική κλίμακα και τεχνολογίες καθαρής καύσης του άνθρακος. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα στην Ευρώπη που να είναι ακριβώς η ίδια τιμή ενέργειας για όλους. Αλλά μέσα στο πακέτο κλιματικής αλλαγής, εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνουμε κάτι για να αντισταθμίσουμε τις δυσκολίες που υφίστανται τα νέα κράτη-μέλη που όπως είπατε εξαρτώνται πάρα πολύ από τον άνθρακα. Δώσαμε <clears throat> για τα υπάρχοντα εργοστάσια που καίνε άνθρακα δωρεάν εκπομπέ κατά κάποιο τρόπο, δωρεάν περιθώρια εκπομπών. προσπαθώντα να μειώσουμε λοιπόν το κόστο που πρέπει να απομισθούν οι πολίτε των χωρών αυτών. Πράγματι, ο άνθρακα θα εξακολουθήσει να είναι μια βασική καυσιμήλη. Επομένω, η τεχνολογία καθαρή καύση είναι καλύτερη από τι παλιέ τεχνολογίε, αλλά ακόμα και οι τεχνολογίε καθαρή καύση άνθρακα θα πρέπει μακροπρόθεσμα να ξεπεραστούν γιατί είναι ρηπαίνουσες, εκπέμπουν διοξίδιο του άνθρακος. Αν βρούμε κάποιες καταπληκτικές τεχνολογίες για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, εντάξει, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να κινόμαστε όλο και πιο προς πιο καθαρούς τρόπους παραγωγής ενέργειας και αγαθών. Πιστεύω επίσης ότι από την οπτική γωνία της ασφάλειας εφοδιασμού ενέργεια θα πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητοι από όλοι. Θα κάψουμε και αυτή θα πρέπει να, αυτό πρέπει να είναι το όραμά μας. Δεν ξέρω αν σας κατάλαβα σωστά. Είπατε ότι στο μέλλον ότι και το, η τεχνολογία καθαρού, καθαρής καύσης άνθρακος και αυτή θα πρέπει να ξεπεραστεί. Είπα ότι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα θα έχουμε τον άνθρακα σαν καύσιμο και στην Ευρώπη. Το γνωρίζω αυτό. Αυτό όμως το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι, ότι στη δική μου μακροπρόθεσμη προοπτική και δεν μιλάμε τα επόμενα πέντε χρόνια θα ήθελα να δω να έχουμε μια κοινωνία με χαμηλή χρήση άνθρακα και μια κοινωνία όπου θα μπορούμε να απεξαρτηθούμε τελείως από τα ορυκτά καύσιμα. Ίσως δεν θα γίνει αυτό στη δικιά σας και τη δική μου ζωή, αλλά μακροπρόθεσμα νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Πάντα ο άνθρωπος μπορεί όταν χρειάζεται να επινοεί τις κατάλληλες τεχνολογίες. Σύμφωνα ο πρόεδρος. Ο Κρήτον έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας καλωσορίζω. Χαίρομαι που βλέπουμε κάποιον που είναι αφιερωμένος στις κλιματικές αλλαγές σε αυτή τη θέση. Θα θέλαμε πάντως και περισσότερη αυτοκριτική για τα σφάλματα της Προεδρίας στην Κοπενχάγη. Στα ελληνικά τώρα. Θα εγγυηθείτε ότι τα φυσικά οικοσυστήματα που είναι οι αποθήκες άνθρακα της γης και εκτελούν ε, την επιτακτικά αναγκή για το πλανήτη απορρόφηση άνθρακα θα προστατευτούν επαρκώς Πιο συγκεκριμένα, πώ θα ενσωματώσετε πολιτικέ για την προστασία του εδάφου, των οικοτόπων, των δασών, των θαλασσών και των υδάτων σε μια συνεκτική πολιτική για την κλιματική αλλαγή, η οποία είναι απαραίτητη τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Uh, we already stressed it a bit with the όλοι ανησυχούμε με αυτήν την πρακτική των παγίδων και μετά το πώς θα υπάρξει η, η γεωργία και η καλλιέργεια των γεών. Πρέπει να έχουμε συντονισμένη θέση στην Ευρώπη. Προς στιγμή δεν έχουμε. Οι γραμμές που ακολουθούμε είναι διαφορετικές, δεν είναι και πολύ βιώσιμες. Δεν γνωρίζουμε το εάν υπάρχει ε, μονιμότητα και διάρκεια και στην δασοκομική μας πολιτική. Πρέπει να συντονιστούμε και θέλω να συνεργαστώ και με τον συνάδελφό μου κύριο Ποτόσνικ με την προϋπόθεση ότι θα με εγκρίνετε ως επίτροπο για να κάνω αυτό που είπατε και εσείς, να δούμε τι γίνεται με τα οικοσυστήματα. Και ε, η, η οδηγία είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για να δούμε την πολιτική μας και την προστασία περιβάλλοντος. Διότι στην οδηγία πλαίσιο για το νερό Τώρα, κάθε κράτος μέλος πρέπει να κάνει τα δικά του εθνικά σχέδια και τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για να δει πώς θα προστατεύσει την, α, τα δάση, τη γη, τα ύδατα και όλα αυτά θα περάσουν μέσα από την οδηγία πλαίσιο για το ύδατο. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί τομεί όπου η, Ένωση τα τελευταία πέντε χρόνια ξεκίνησε με πολύ σημαντικές οδηγίες υπό την αιγίδα του κυρίου Δήμα και νομίζω ότι πρέπει να συνεργαστούμε και να τα εφαρμόσουμε όλα αυτά έτσι ώστε να μας βοηθήσουν όλα αυτά για να εκπληρώσουμε το στόχο μας να είμαστε περισσότερο βιώσιμοι. Ποια μέτρα σκοπεύετε να πάρετε προκειμένου να διασφαλίσετε ότι η προστασία των τροπικών δασών δεν θα καταλήξει να γίνει ένας τρόπος αντιστάθμισης εκπομπών αερίων, αλλά θα αποτελεί ανεξάρτητο πυλώνα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Συμφωνείτε πως οι δεσμεύσει μείωση εκπομπών θα πρέπει να μεταφράζονται σε πραγματικέ μετρήσιμε μειώσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αν ναι, πώ σκοπεύετε να το πετύχετε. This question about tropical... Για το θέμα των τροπικών δασών και το πώς πρέπει να φροντίσουμε να μην καταλήξει απλώς ως αντισταθμιστικό μηχανισμός. Ένα εργαλείο θα ήταν να έχουμε ξεκάθαρους κανόνες διεθνώς ως τμήμα διεθνούς συμφωνίες. Να μην προσμετρήσουμε διπλά τα δάση αυτά παραδείγματος χάρη και τελικά να έχουμε μια, ένα σωστό αντάλλαγμα για τα χρήματά μας. Δηλαδή να μην κατά κάποιο τρόπο συμπεριλάβουμε δασοκομικά μέτρα τα οποία ούτως ή άλλως θα λάμβαναν χώρα. Δηλαδή πρακτικές που ήδη συμβαίνουν να μην προσμετρηθούν ως κλιματική ε, ε, δράση. Όχι, διότι αυτό θα το κάνατε ούτως ή άλλως. Θα πρέπει δηλαδή να προσμετρηθούν μόνο τα επιπρόσθετα πράγματα που κάνετε στη δασοκομική σας πολιτική. Μόνο αυτό θα πρέπει να προσμετρηθεί στην κλιματική σας προσπάθεια. Αυτό είναι ένας από τους πολύ δύσκολους τομείς και στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, αλλά είναι επίσης και ένας τομέας όπου έχουν το περισσότερο προοδεύσει ή διαπραγματεύσεις και έτσι να βοηθήσουμε να, τον Γεωργό στην αναπτυσσόμενη χώρα εκεί που προστατεύει το δάσος και δεν το καταστρέφει και να του δώσουμε μια χρηματική ε, αντιστάθμιση και εμείς να, να τον αφήσουμε να διατηρήσει εκεί αυτό το δάσος. Επόμενη ερώτηση, ερώτηση κυρία Καθλίν Φαντ Ε, εδώ είμαι, εδώ είμαι κυρία Υπουργέ. Ε, γεια σας και καλώς ήλθατε. Έχει περάσει το 50% του χρόνου α, της ακρόασης και σε γενικές γραμμές με πείθετε για τις ικανότητές σας. Όμως το χαρτοφυλάκιό σας μοιάζει λίγο αδύναμο, γιατί θα πρέπει να σας ελεήσουν άλλα χαρτοφυλάκια, άλλοι επίτροποι, για να αυξήσετε τα κονδύλια σας. Αφού αυτά που είπε η Μπρίτα Τόμψον, ας πούμε, τι είσαστε, ε, ε, είσαστε έτοιμοι να, να κάνετε μια συντονισμένη προσπάθεια για όλες τις επιδοτήσεις προκειμένου να αποστασιοποιηθούμε από τα ορυκτά καύσιμα και την πυρηνική ενέργεια. Μιλάω για τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, ε, γιατί νομίζω ότι ο, ένας επίτροπος για το κλίμα αυτή τη στάση πρέπει να έχει. Φυσικά, θα ήθελα οι πόροι να πηγαίνουν προς μια κατεύθυνση ε, επωφελή για το κλίμα. Το είπα ξεκάθαρα ότι δεν θέλω οι επιδοτήσεις ε, να πηγαίνουν στα ορυκτά καύσιμα ούτε στην Ευρώπη αλλά ούτε και αλλού. Αν είσαι φυσικά Ινδονήσιος και φτωχός, ε, θεωρείς ότι αυτό είναι και κοινωνική πολιτική. Αλλά και τώρα, ακόμα και η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας δεν συστήνει τις επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα. Δεν πρέπει να τις δίνουμε, δεν θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκή πολιτική. Τώρα, έχετε δίκιο ότι ότι η γενική μου διεύθυνση και όσα είπατε για αυτήν ισχύουν. Δεν θα είναι πολύ εύκολο να αναπτύξω μια στρατηγική. Και κάποιοι από εσά ξέρω ότι έχουν ανησυχίες και αβεβαιότητες για το χαρτοφυλάκιό μου. Η σημερινή μας συζήτηση αποδεικνύει ότι το κλίμα μπορεί να είναι τα πάντα. Βιομηχανία, ανάπτυξη, έρευνα, περιβάλλον, ενέργεια, μεταφορές είναι σαφές ότι πρέπει να κάνουμε βαθιές επιλογές. Ε, γιατί όλα αυτά δεν μπορούμε να τα προωθήσουμε παράλληλα. Ε, θα πρέπει να το κάνουμε αντίθετα. Το κλίμα το βάλουμε σε όλες τις πολιτικές. Φυσικά είναι σαφές ότι έχουμε εργαλεία για να το εντάξουμε σε άλλες πολιτικές. Ε, και επίσης είναι σαφές ότι όταν η Επιτροπή λέει ότι θα δώσει μεγάλη προτεραιότητα στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και ότι θέλει να εντάξει το κλίμα σε όλες τις πολιτικές, το λένε όλα τα έγγραφα της Επιτροπής αυτό, ε, τότε σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να εξοικονομήσουμε και τους απαραίτητους πόρους, ούτως ώστε αυτό να γίνει. Η κυρία Κορχόλα. Η κυρία Κορχόλα, κυρία υποψήφια επίτροπε, έχετε εκφράσει την πεποίθησή σας ότι θα λειτουργεί το σύστημα εμπορία εκπομπών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλετε να το συνδέσετε με άλλα εξίσου ε, ευέλικτα συστήματα σε άλλες χώρες έξω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό περιλαμβάνει όμως και ποσά ε, και εκπομπές κατά χωρίς κόστος. Ξέρουμε ότι ακριβώς το πόσο πολλές είναι αυτές οι εξαιρέσεις, οι τα πιστοποιητικά που παίρνει κανεί σε μηδενική αξία είναι αυτά που καθορίζουν την αξία των πιστοποιητικών στην ευρύτερη αγορά. Ποια είναι τα όρια που θέλετε να θέσετε λοιπόν. Το Κογκρέσιο των ΗΠΑ συζητά την ελάχιστη και τη μέγιστη τιμή των πιστοποιητικών. Δεν έχουμε τέτοια ρύθμιση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με ποιο τρόπο θα συνδέσετε λοιπόν δύο συστήματα τα οποία έχουν και βασίζονται και σε διαφορετικά νομίσματα εξάλλου από ό,τι κατανοώ, δεν είναι απαραίτητο να έχουμε ακριβώς τα ίδια πιστοποιητικά σε όλα τα μέρη του κόσμου. Θα ήταν όμως εποφελές αν μπορούσαμε να θέσουμε κάποια πρότυπα. αυτός είναι ο ευρωπαϊκό τρόπος με τον οποίο κάνουμε τα πράγματα. Να υπάρξει ένα πρότυπο το οποίο θα ακολουθηθεί και από τους άλλους. Αυτό θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Αν θα μπορούσαμε λοιπόν να επιτύχουμε μια σύνδεση μεταξύ του ευρωπαϊκού συστήματος και του αμερικανικού συστήματος το οποίο θα εφαρμοστεί τώρα, θα έχαμε εξασφαλίσει ότι αυτά τα συστήματα, το κοινό αυτό σύστημα θα μπορούσε να υιοθετηθεί και από άλλες χώρες, από την Αυστραλία, την Ισλανδία, ε, την Ιαπωνία. Φυσικά, το... ο στόχος μας θα πρέπει να είναι να έχουμε ένα παγκόσμιο σύστημα με παγκόσμια τιμή άνθρακος. Γι' αυτό Πιστεύω ότι θα ήταν προτιμητέο <clears throat> και βέλτιστο στην Ευρώπη να μην έχουμε διαφορετικά συστήματα, 27 διαφορετικά συστήματα πληστηριασμού πιστοποιητικών εκπομπών. Να γίνει με ένα κεντρικό τρόπο, να γίνεται η διαδικασία πληστηριασμού στην Ευρώπη και η Ευρώπη να αναλάβει την πλήρη κατανομή των πιστοποιητικών εκπομπών. Αυτό είναι ο πιο ισχυρό τρόπο να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Αυτό το οποίο βέβαια είναι η ανησυχία πολλών είναι ότι υπάρχει ευρεία ε, κερδοσκοπία στις ε, χρηματαγορές και τα hedge funds ίσως θα θελήσουν να μπουν σε αυτή την αγορά. Επομένως είναι απαραίτητο να υπάρχει και κάποια καλύτερη μορφή σχεδιασμού στον τομέα αυτό, λέει ο Πρόεδρος. Αυτή ήταν δική μου παρατήρηση. Ακολουθεί η Φιώνα Χόλ στο επόμενο ερώτημα. Γι' αυτό ακριβώς το θέμα στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίων Εγκουπομπών υπήρξε ένα πρόβλημα. Γιατί για να δουλέψει το σύστημα πρέπει να έχετε μια σταθερή και αυξανόμενη τιμή για τον άνθρακα. Και για διάφορους λόγους. Πρακτικά υπάρχει και η οικονομική κρίση αλλά και τα λοιπά. Η τιμή λοιπόν του άνθρακα ήταν ασταθής και αδύναμη. Συμφωνείτε με την επιβολή ελάχιστης τιμής για τον άνθρακα τουλάχιστον ως βραχυπρόθεσμο μέτρο. Απάντηση. Η ιδέα αυτή συζητείται και διεθνώς και στην Ευρώπη εδώ και καιρό και το συζητούν και στις ΗΠΑ. Αμφιβάλλω το εάν θα βοηθήσει αυτό τα όσα προσπαθούμε να επιτύχουμε. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Δηλαδή αν έχετε αυτή την ελάχιστη τιμή, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι στην επόμενο οικονομικό κύκλο δεν θα υπάρξει και αίτηση για μέγιστη τιμή. Οπότε στην ουσία, στο τέλος, θα έχετε πάλι ένα πολύ παρεμβατικό σύστημα. Ξέρω ότι καλό θα ήταν, λένε ορισμένοι καλό θα ήταν να έχουμε μια ελάχιστη τιμή, αλλά μην ξεχνάμε ότι από ό,τι καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή η τιμή διακυμαίνεται ανάμεσα στα 10 και 25 ευρώ. Σε σύγκριση με τη διακύμανση του πετρελαίου, της τιμής του πετρελαίου, δεν είναι και τόσο μεγάλη αυτή η διακύμαση. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πιο σημαντικό να είμαστε πολύ καλοί στο να μην δώσουμε πολλά δωρεάν δικαιώματα εκπομπών. Εκεί πρέπει να γίνει ο έλεγχος και μετά ας δουλέψει μόνη της η αγορά. Βλέπω πολλές περιπλοκές εάν ξεκινήσουμε αυτήν την ελάχιστη τιμή και αν υπάρχει πλεόνασμα των δικαιωμάτων εμείς θα τα αγοράσουμε τι να σας πω, φαίνεται ναι μεν ελκυστικό γιατί όλοι θέλουμε να έχουμε αυτήν την προβλεπτικότητα, αλλά φοβάμαι τι θα συμβεί όταν η βιομηχανία έρθει μετά και μας πει και τώρα θέλουμε μέγιστη τιμή. Τι θα κάνουμε, θα έχουμε μετά καθορισμένη τιμή, πώς θα δουλέψει μετά η, αγορά. Το ότι οι τιμές μειώνονται σε περίοδο κρίσης δεν είναι και τόσο δύσκολο να το μαντέψει κανένας. Δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση, κατεβαίνουν οι τιμές. Οπότε εμπιστευόμαστε την αγορά ότι θα τα καταφέρει μόνη της. Κυρία Καβάλιο. Η e έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη των καθαρών τεχνολογιών είναι ένας βασικός πυλώνας αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Στον τομέα της ενέργειας η Ευρώπη έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια λιγότερο από ό,τι στη δεκαετία του 1980. Πώς θα εξασφαλίσετε ότι οι μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές θα υπάρξει πραγματική επένδυση για τα θέματα αυτά. Και σε ό,τι αφορά την ε, ευρωπαϊκή ικανότητα παραγωγής καθαρής ενέργειας, ηλιακής ενέργειας, των εφιών δικτύων, πώς θα αναπτύξετε αυτές τις ε, κατευθύνσεις. Θα έχετε θα υπάρξει υπάρχουν προγράμματα για τη μείωση των εκπομπών στις πόλεις με συμμετοχή των Δημοτικών Συμβουλίων. Πώς θα δώσετε την, ε, και κίνητρα για την ε, αποτελεσματικότητα της ενέργειας στα κτίρια και την μικροπαραγωγή ενέργειας. the... Μιλήσατε για τα κτίρια, μιλήσατε για την έρευνα, εντάξει. Είναι κεφαλαιώδες όταν κάνουμε μια συζήτηση για τις δημοσιονομικές προοπτικές, όπως το είπα και προηγουμένως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να θεσπίσουμε τις προτεραιότητες μέσα στις δημοσιονομικές προοπτικές σωστά γιατί πρέπει να συντεριάζονται με τις πολιτικές μας προτεραιότητες. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τις ίδιες προοπτικές τα επόμενα πέντε χρόνια όπως τα προηγούμενα πέντε χρόνια. Γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε καινούργιε ιδέε. Κάποια πράγματα θέλουμε να τα κάνουμε διαφορετικά. Και ένα από του τομεί όπου πρέπει να δώσουμε έμφαση και έχετε μεγάλο δίκιο. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί κάπω η χρηματοδότηση της έρευνας σε μερικά τουλάχιστον κράτη-μέλη <clears throat> και με το πρόγραμμα οικονομικής ανάκαμψης δίδεται προτεραιότητα στην έρευνα για τις ανανεώσιμες ενέργειες αλλά η μακροπρόθεσμη πορεία ήταν η μείωση των επενδύσεων στον τομέα αυτό και αυτό δεν είναι ιδιαίτερα σόφρον πολιτική αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα ισχυρά σημεία της Ευρώπης. Η Ευρώπη έχει μεγάλη ικανότητα στον τομέα αυτό και όταν πρόκειται τώρα για ταμεία για τη γεωργία και εκεί θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερα ποσά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για έρευνα νέε τεχνολογίε για την παραγωγή φυσικού αερίου από τη γεωργία παραδείγματο χάρη. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό νέο μια νέα σημαντική οδό. Δεν πρέπει να περιμένουμε από όλα τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν αυτήν την οδό. Θα πρέπει καταρχήν να πιέσουμε να γίνει αυτό από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουμε ένα πιο καθαρό περιβάλλον. Είναι σημαντικό λοιπόν να αγωνιστούμε μέσα στου διάφορου τομεί να υπάρξει μεγαλύτερη χρηματοδότηση της έρευνας. Αν εγκριθώ από εσά ε, ως Επίτροπος για την κλιματική αλλαγή, αυτό θα είναι μία από τις πρώτες επαφές που θα ένα από τα πρώτα θέματα που θα έχω σε επαφέ με τον συνάδελφό μου, τον Επίτροπο Έρευνα, γιατί θα προσπαθήσουμε να δούμε πώ μπορούμε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σάιντερ Καντράουι, από την Επιτροπή Μεταφορών. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ είμαι. Σας γνέφω, κύριε Επίτροπε, υποψήφια Επίτροπε. Τονίσατε τη σημασία των μεταφορών στην ε, συζήτηση για το κλίμα. Φυσικά έχει τη μερίδα του λέοντος τις ε, εκπομπές. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε μέτρα για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. δεν θα πρέπει τα ελαφρά εμπορικά ας πούμε, οχήματα να έχουν δικό τους ε, ποσοστό για τις εκπομπές. Μιλήσατε για το κλιματικό πακέτο. Τι χρονοδιάγραμμα έχετε στο μυαλό σας. Θα μπορούσατε να είστε πιο συγκεκριμένοι για την δική σας άποψη, για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις μεταφορές από την άποψη του κλίματος. Η απάντηση είναι το, το συντομότερο δυνατόν για το χρονοδιάγραμμα που με ρωτήσατε. Αλλά φυσικά θα πρέπει να το συζητήσω και με τον Επίτροπο για τις μεταφορές. Αυτό. Νομίζω ότι έχουμε μια τεράστια πρόκληση με τις εκπομπές από τις μεταφορές που αντισταθμίζουν οτιδήποτε κάνουμε, οτιδήποτε επιτυγχάνουμε σε άλλους τομείς. Ε, επίσης, αν αλλάξουμε τα πράγματα, παραδείγματος χάρη στους σιδηροδρόμους, χρειάζεται παραπάνω από πέντε χρόνια, χρειάζονται δέκα χρόνια. Από τη στιγμή που αποφασίζουμε να κάνουμε κάτι μέχρι να έχουμε αυτά αποτελέσματα. Γι' αυτό λοιπόν ε, το θέμα επήγει. Σας είπα προηγουμένως ε, ότι για τα φορτηγά θα πρέπει να είναι μία από τις πρωτοβουλίες. Θα πρέπει να, έχουμε, να αναθεωρήσουμε το εργαλείο που έχουμε στην Ευρώπη ε, Επίση, ανέφερα την αυσιπλοεία. Θα πρέπει να συμπεριλάβουμε την αυσιπλοεία, αλλά εγώ και ο Επίτροπο Μεταφορών θα πρέπει να δούμε συνολικά τον τομέα των μεταφορών. Θα, γιατί τα πράγματα αυτά είναι αλλοσυνδεδεμένα. Και στο μάτι του πολίτη, αν οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν ε, τα τρένα για τις δημόσιες μεταφορές, φταίμε κι εμείς θα πρέπει να μοιραστούμε τι βέλτιστε πρακτικέ. Ξέρω ότι πολλά από τα θέματα, παραδείγματο χάρη σχεδιασμό, ε, είναι θέμα των κρατών μελών. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει ε, να διαδώσουμε με καλύτερο τρόπο, πιο αποτελεσματικά, τι τις ε, βέλτιστε μεταφορέ. πέρυσι στη Δανία είχαμε ένα τεράστιο σχέδιο μεταφορών για πρώτη φορά. Ένα επενδυτικό σχέδιο και προσπαθούμε να δούμε με πρακτικό τρόπο πώς θα εξασφαλίσουμε επιδοτήσεις. Ε, τα δύο τρίτα των επενδύσεων αυτών θα πάνε στις δημόσιες μεταφορές. Ε, πολλά μπορούμε να κάνουμε για την ηλεκτροδότηση, φυσικά με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Και με αυτόν τον τρόπο ε, μπορούμε και εκεί να βοηθήσουμε με τον καθορισμό προτύπων. Ε, σας ευχαριστώ για την απάντησή σας. Να πάω τώρα σε ένα άλλο σημείο που συνδέεται όμως με τα προηγούμενα. Στον τομέα των μεταφορών εδώ και χρόνια γίνεται μια συζήτηση για την τιμολόγηση. Προσπαθούμε να το βοηθήσουμε τον κόσμο να αλλάξει συμπεριφορά μέσω της εσωτερήκευσης του εξωτερικού κόστους. Και το ε, του άνθρακα είναι ένα σημαντικό εξωτερικό κόστος, ένα από τα πολλά, αλλά σημαντικό. Εσείς υποστηρίζετε αυτή την έννοια, αυτή την αρχή της εσωτερικοποίησης του εξωτερικού Κόστου τις μεταφορές. Και ποιο εργαλείο είναι το καταλληλότερο για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Ναι, το υποστηρίζω και είναι σημαντικό να, είμαστε, να έχουμε ανοιχτό πνεύμα και να υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Φυσικά, ουσιαστικά είναι φορολόγηση και οικονομικό θέμα και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποφασίσουν να το χρησιμοποιήσουν, πώς θα το χρησιμοποιήσουν κτλ. Αλλά η εσωτερήκευση του εξωτερικού κόστους είναι ένα κατάλληλο εργαλείο. Μερικές από τις αλλαγές που θα πρέπει να περάσουν σε αυτόν τον τομέα ε, γίνονται, αν σκεφτούμε, πιο εφάνταστα, λιγότερο συμβατικά. Παραδείγματο χάρη, ο κόσμος θα πρέπει να πληρώσει για κάποιες ε, ώρες της ημέρας αν θέλει να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό του, Φερρυπίν. Ε, φυσικά θα πρέπει να, χτίσουμε, να φτιάξουμε και δρόμους. Α, αλλά δεν θα πρέπει να φτιάχνουμε δρόμους ε, οι οποίοι φτιάχνονται για να χρησιμοποιηθούν μία-δύο ώρες της ημέρας, ας πούμε. Ε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και την τεχνολογία και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και την, α, τις τιμές. Κάποιοι θα πρέπει να πληρώνουν για, κάποιους, ε, για κάποιες υπηρεσίες. Πάμε στον πέπτο γύρο. Ο πρώτος είναι ο κύριος Ρόντε. Μάλιστα. Ακούσαμε πολλά αυτή την εβδομάδα. Πιστεύω ότι η επίδοση σας είναι όμως πολύ καλή. Ακούσαμε ακροάσεις και υποψήφιους επιτρόπους με πολύ ισχυρή προσωπικότητα όπως ο κ. Ζέτιγκερ του οποίου ίσως είναι λίγο διαφορετική η θέση. Ο υποψήφιος επίτροπος για θέματα έρευνας δεν θέλει να χρησιμοποιήσει ούτε ένα ευρώ από την έρευνα για την πυρηνική ενέργεια για άλλους σκοπούς και μετά ακούσαμε και τα όσα αναφέρθηκαν για τις ε, γεωργικές επιδοτήσεις. Πώς θα πείσετε τους συναδέλφους σας να μεταφέρουν τις αρμοδιότητες τους από τα δικά τους χαρτοφυλάκια στο δικό σας. Πώς θα ε, εξασφαλίσετε την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ξέρω ότι θα πρέπει κανένας να δώσει μάχη. Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Αν πάτε σε ένα συνάδελφο και του πείτε ότι πρέπει να σκεφτείς και την κλιματική διάσταση ενώ αυτός ο συνάδελφος έχει και άλλες δέκα προτεραιότητες να λάβει υπόψη του θα δοθεί μία μάχη αλλά κοιτάξτε συνολικά την Κομισιόν δεν είναι ε, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος ή, ο Επίτροπος ε, Ενέργειας μόνο πρέπει όλοι οι Επίτροποι να μεταφράσουμε τα λόγια μας σε έργα και αυτά θα πρέπει να τα κρίνουμε σε πέντε χρόνια εγώ πιστεύω ότι είναι δυνατόν να υπάρξει βάσιμη επιχειρηματολογία και όσοι είναι υπεύθυνοι για την καινοτομία, για την πρόθεση της απασχόλησης, για την πρόθεση της βιομηχανίας, όχι μόνο σε 5 αλλά σε 10-20 χρόνια να δουν τα ωφέλη. Δεν θα είμαι απομονωμένη και μόνο μου. Θα πρέπει να συνεργαστώ σε στενή ε, θα, θα, θα εργαστώ σε στενή συνεργασία με τους συναδέλφους και θα προσπαθήσω να παρουσιάσω την ε, θέση μας. Και ο γενικός μου διευθυντής έχει μεγάλη εμπειρία και θα πρέπει να με βοηθήσει να παρουσιάσω ισχυρά επιχειρήματα προς όφελος όλων μας. Ευχαριστώ. Κάποιος από τους μη εγγεγραμμένους είναι εδώ για να θέσει ένα ερώτημα. Όχι. Δεν έχουν παραστεί λοιπόν στην ε, ακρόαση. Το επόμενο ερώτημα στην Judith Μέρκες. Ευχαριστώ. Είμαι εδώ στα αριστερά σας. Κύριε Χέντεγκάρτ, η Κοπενχάγη δεν απέδωσε τα προσδοκόμενα αποτελέσματα και εσείς φυσικά που περιμένατε. Όπως αναφέρατε, μία λύση για τα προβλήματα αυτά είναι να μιλάει η Ευρώπη με μία ενιαία φωνή και εσείς φαίνεστε αποφασιστικοί και πεπισμένοι ότι αυτό είναι απαραίτητο. Μπορώ να υποθέσω λοιπόν ότι θα δεσμευτείτε για να προσπαθήσετε να πείσετε την Κομισιόν, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για να προχωρήσουμε το θέμα, να προχωρήσουμε αυτό το θέμα και να το κάνουμε μια πραγματικά ε, ε μοναδική, αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μια μοιραζόμενη με τα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι η συνθήκη της Λισαβόνας κάνει σαφές ότι θα υπάρξει ένας διαπραγματευτής από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη η συνθήκη της Λισαβόνας αντιμετωπίζει το θέμα αυτό, ότι υπάρχει ένας, κύριο κύριος διαπραγματευτής και αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει πολύ σύντομα. Ίσως γίνεται σήμερα και αύριο στη Σεβίγια, στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος. Γιατί ακόμα Πάρα πολλοί έχουν μείνει στην Κοπενχάγη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να σκεφτούμε ότι το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Φεβρουάριο θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει τα θέματα αυτά. Δεν είναι εύκολο βέβαια να αποφασίσουμε ποιο θα πρέπει να κάνει, θα πρέπει να αναλάβει να είναι ο διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να υπάρξουν διαμάχες, αλλά οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από πολλά χρόνια έχουν ήδη κατανοήσει πώς λειτουργεί ο θεσμικός μηχανισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουν να δουν την Ευρώπη να λειτουργεί με πιο ενιαίο τρόπο και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να ξασφαλίσω ότι θα ακουστεί η δική μου φωνή στο Συμβούλιο όταν έχω την ευκαιρία να είμαι στο Συμβούλιο και μέσα στην Κομισιόν, γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα και τον πρόεδρο τη Επιτροπής μετά από ένα ενημερωτικό ερώτημα. Στην, ε, μέχρι την 31η Ιανουαρίου, ποιος ε, διατυπώνει αυτές τις δεσμεύσεις, τα κράτη-μέλη και τα 27 ή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να συζητηθεί αν κατάλαβα καλά. Θα... Την επόμενη εβδομάδα θα συζητηθεί στο Κορεπέρ. Συζητήθηκε και αυτή η εβδομάδα, μάλιστα. Και από ό,τι μου είπαν, θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις από τα κράτη-μέλη. Εγώ νομίζω ότι είναι λογικό η Ευρώπη να έχει ένα νούμερο, όπως κάναμε και στο Κιώτο, να δώσει, να δεσμευτεί ως προς ένα νούμερο και συνεχεία μπορούμε να δούμε τι ποσοστό αναλογεί στο κάθε κράτος μέλος. Αλλά αυτό είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να γίνει πριν την 1η Φεβρουαρίου. Και επομενω πριν αναλάβω τη θέση του Επιτρόπου, αν την αναλάβω. Χειροκρότησα, γιατί συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπατε. Η μόνη φορά που συμφωνήσατε ήταν αυτή, δηλαδή. Μόνο εγώ χειροκρότησα, αλλά νομίζω ότι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι στην πραγματικότητα συμφωνούν με αυτή τη θέση. Γιάννικ Ζαντό. Κυρία Επίτροπε, υποψήφια Επίτροπε, αναφερθήκατε στις διαφορές μεταξύ κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω ότι στη Γερμανία, στη Γαλλία και στη Βρετανία αυτό το μήνυμα θα το ακούσουν οι ηγέτες. Αλλά τις διαφορές στο εσωτερικό της Επιτροπής πώς θα τη διαχειριστείτε. Συχνά ε, ο λόγος σας είναι αμφίσιμος, ειδικά για το στόχο 30%. Λέτε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να παίξει ηγετικό ρόλο, ότι άλλες χώρες όπως η Κίνα κινήθηκαν και άλλαξαν στάση, αλλά ταυτόχρονα λέτε ότι αν δεν τα καταφέρουν, δεν θα τα καταφέρουμε κι εμείς, θα πρέπει να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις, αλλά δεν είναι κατάλληλη στιγμή. Δεν καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο στόχος σας, ο δικός σας στόχος. Επίσης, στο εσωτερικό των υπηρεσιών σας, τι ρόλο θα παίξετε για τη συζήτηση για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Συχνά, ε, για το θέμα των αγορών του άνθρακα υπάρχει πρόβλημα. Και τελικά δεν προωθούμε μια αφιλόδοξη ενεργειακή πολιτική. Τελικά, πέστε μας, θα προωθήσετε ένα δεσμευτικό στόχο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στην Ευρώπη. Πέρα από την, τα θεληματικά σας λόγια θα προωθήσετε αυτή την πρωτοβουλία, δηλαδή έναν δεσμευτικό στόχο για την ενεργειακή απόδοση. Νομίζω ότι για Έχουμε ήδη για, τα, για τις ανανεώσιμες ενέργειες και για τις εκπομπές έχουμε δεσμευτικούς στόχους. Το 20% σας στόχος για την ενεργειακή απόδοση είναι και αυτό μια πρόταση η οποία έχει τεθεί. Δεν χρειάζεται να είναι δεσμευτικός όμως ο τελευταίος στόχος, <clears throat> γιατί αν θέλουμε να το κάνουμε αυτό, τότε τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εστιάσουν πάρα πολύ στην ενεργειακή απόδοση και δεν θα μπορέσουν να επιτύχουν τους άλλους στόχους. Ξέρουμε ότι συζητήθηκε πάρα πολύ αυτό το θέμα κατά τη διάρκεια της συζήτησης του πακέτου κλίματος και ενέργειας και δεν νομίζω ότι έχει νόημα να επαναλάβουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί τα επιχειρήματα θα παραμείνουν τα ίδια. Θα έλεγα για το 30%, την επίτευξη του 30%. Δεν νομίζω ότι λέω διαφορετικά πράγματα κατά καιρού. Εγώ έχω υποστηρίξει πάντα το να προχωρήσει η Ευρώπη στο 30%. Ήμουνα πάντα υπέρμαχος αυτής της άποψης. Απλώς αυτό το οποίο είπα προηγουμένως σήμερα το πρωί είναι ότι βλέποντας τα πράγματα εκ των υστέρων βλέποντας τι έγινε αυτό στην Κοπεχάγη που η Ευρώπη δεν πέτυχε το 30%. <laughs> δεν μπορώ να σας ρωτήσω, αλλά μήπως θα συμφωνούσατε κι εσείς ότι θα ήταν καλύτερο να κρατήσουμε το 20% με την δυνατότητα να φτάσουμε στο 30% εν καιρό για να δούμε αν θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε κάποια, να επιτύχουμε κάτι περισσότερο σε επίπεδο ποσοστό από τους άλλους εταίρους μας. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να συζητάμε το τι θα είχε γίνει αν η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε άλλη στρατηγική πριν από την Κοπεχάγια. Βλέποντας τα πράγματα όπως είναι τώρα, δεν θα είναι καλύτερο να έχουμε αυτήν την δυνητική στάση σε τακτικό επίπεδο. Νομίζω ότι από αυτά τα οποία έχω ακούσει στην Κοπεχάγη και στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος αν ξανανοίξουμε τώρα αυτή τη συζήτηση δεν πρέπει να αυταπατώμεθα. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να μην συμφωνήσουμε πια στο 30%. Σπίνιερ τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Πολωνία έχει μεγάλη θέση στις εκπομπές του θερμοκηπίου και σύμφωνα με τη συμφωνία του Κιώτο χρειάστηκε μείωση 60 και 30% και θα πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι οι, οι χώρες των τα προηγούμενα κράτη-μέλη, τα 15 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους έπρεπε να είχαν εκπληρώσει μεγαλύτερες. Οπότε δεν είναι τώρα υποκριτικό να ζητήσουμε από τα νέα κράτη να αναλάβουν αυτό το μεγάλο βάρος εξαιτίας της πολιτικής αυτής. αυτού του είδους η πολιτική σημαίνει ότι οι φτωχότερες χώρες της Ένωσης στην ουσία θα επιδοτήσουν τις πιο πλούσιες χώρες και κράτη-μέλη. Πώς το βλέπετε αυτό σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Συνοχή. Δεν κατάλαβα ακριβώς τη μετάφραση, αλλά για το ποιος κάνει τι. Όταν κάναμε το πακέτο ενέργειας και κλίματος, Ορισμένοι από εμά θα ήθελαν πληστηριασμού 100% το ταχύτερο δυνατόν. Κάποιοι δεν το ήθελαν. Νομίζω ότι βρέθηκε ένα συμβιβασμό, ο οποίο κατά κάποιο τρόπο αντιστάθμισε τα νέα κράτη-μέλη με δωρεάν παροχές για τα υφιστάμενες μονάδες παραγωγής ενέργειας. Το είπατε κι εσείς. Και τώρα για τις νέες κατασκευές, τότε εκεί πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι ίση όροι για όλους. Γιατί αλλιώς ορισμένοι απλώς θα κατασκευάσουν μια μονάδα παραγωγής ενέργειας σε ένα άλλο κράτος μέλος γιατί σε αυτό το κράτος μέλος έχετε δωρεάν εκπομπές, στο άλλο όχι. Δεν νομίζω ότι δικαιολογείται αυτό. Äh, ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λίχτεμπεργκ, ευχαριστώ πολύ. Εδώ είμαι. Είναι ενθαρρυντικό φυσικά αυτό το οποίο λέτε, ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα των μεταφορών. Γιατί είναι μεγάλη οι ρυθμοί αύξηση ε, στον τομέα των μεταφορών που μπορούν να ακυρώσουν όλες τις πρόοδους στους άλλους τομείς. Βέβαια έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ ισχυρά λόμπι στον τομέα της μεταφοράς, είτε πρόκειται για τις αεροπορικές μεταφορές, είτε πρόκειται για την, ε, τις θαλάσσιες μεταφορές. Παραδείγματο χάρη το θέμα τη ε, απελευθέρωση από την, της από επιδοτήσει ήταν πολύ δύσκολο. Εσείς πού βλέπετε τώρα τι δυνατότητε να υπάρξουν στρατηγικέ πρόοδοι στον τομέα των μεταφορών και πώς θα αντιμετωπίσετε θέματα όπως η σύμβαση των Άλπαιων με τους περιορισμούς που επιβάλλει, μηχανισμούς λοιπόν που μπορούν να είναι εργαλεία για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα πάντα στην πολιτική κλίματος στον τομέα των μεταφορών. Εγώ ήδη δεν μπορώ να πω ότι γνωρίζω τις λεπτομέρειες της ε, Αλπικής Σύμβασης. Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε το συγκεκριμένο αυτό θέμα. Αλλά νομίζω ότι αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Ότι υπάρχει πραγματικά, υπάρχουν πολύ ισχυρέ ομάδες πιέσεων στον τομέα των μεταφορών. Και όταν προσπαθούσαμε να επιτύχουμε τους στόχους για τις εκπομπές των αυτοκινήτων, οχημάτων, ήταν πολύ ισχυρό το λόμπι και μερικές φορές βλέπω τι είδους ε, επιστολές παίρνουμε. Παίρνω ακόμα και σαν υποψήφια επίτροπος πόσο μεγάλη πίεση ασκείται από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Εγώ πάντα είμαι έτοιμη να ακούσω τα επιχειρήματα όλων. Νομίζω ότι είναι πιο ενδιαφέρον να ακούσουμε αυτά που λένε τα λόμπι, που πολλές φορές έρχονται με εναλλακτικές λύσεις για να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα αντί να λένε ότι κάποιος άλλος θα πρέπει να λύσει το πρόβλημα. Έρχομαι βέβαια από το μικρό βασίλειο <laughs> της ε, Δανημαρκίας και αυτός είναι ένα νέος κόσμος, το λόμπι στον οποίο πρέπει να μπω. Υπάρχουν πολλά καλά πράγματα στην Σύμβαση των Άλπαιων, αν θέλετε να, τα, να την διαβάσετε, λέει ο πρόεδρος. Έκτη και τελευταία ομάδα ερωτήσεων και δίνω καταρχήν το λόγο στο Μάρτιν Κάλαναν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν σας επιβεβαιώσουμε και σας δεχτούμε ως ε, ε, Επίτροπος, ένα από τα καλά από τη δουλειά θα είναι το υπηρεσιακό αυτοκίνητο. Θα υποφεληθείτε από αυτό το προνόμιο και τι όχημα θα επιλέξετε για να σας μεταφέρει στις προσωπικές σας διαδρομές. Όταν είσαι υποψήφιος επίτροπος και πρέπει να περάσεις από αυτήν την ανάκριση των τριών ωρών, δεν σκέφτεσαι τέτοια πράγματα, τι αυτοκίνητο θα επιλέξεις κτλ. Τα έχω αφήσει για αργότερα. Ως ε, υπουργό ε, Κλίματος και Ενέργειας και τώρα ως Επίτροπος Περιβάλλοντος, ε, σίγουρα θα διαλέξω το καλύτερο δυνατό ενεργειακά αυτοκίνητο που υπάρχει στην αγορά. Το ίδιο θα κάνω και για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο. Είναι φυσικό και πιστεύω ότι είναι σημαντικό. Όσοι από εμάς έχουμε διαφορετικές θέσεις, να αποδείξουμε στους ε, πολίτες ότι αυτά που λέμε τα εννοούμε. Και να είμαστε ευσυνείδητοι και στην καθημερινότητά μας. Ήξερα θα, το αποφύγετε, θα την αποφύγετε την ερώτηση σας. είναι άλλη μια ευκαιρία. Θα διαλέξετε υβριδικό, ηλεκτρικό, ευρωπαϊκό αυτοκίνητο με βιοκαύσιμα. Και όταν ήσασταν υπουργό στη Δανία είχατε την ίδια ευκαιρία. Ε, τι αυτοκίνητο διαλέξατε στη Δανία. όλε τι άλλε ερωτήσει απαντήσατε. Α, με προκαλείτε τώρα. με προκαλείτε να πω κάτι άσχημο για κάποια αυτοβιομηχαν... αυ... αυτοκινητοβιομηχανία, τη μία ή την άλλη. Εμεί στην Δανία δεν παράγουμε καθόλου αυτοκίνητα. Και επομένω δεν θα πάρω δανέζικο αυτοκίνητο, δεν υπάρχει. Θα πάρω το καλύτερο αυτοκίνητο σε ό,τι αφορά τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα και σε ό,τι αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητά του. Για να δούμε ποιος θα κερδίσει τη μάχη. Χρειάζομαι ένα-δύο μήνες για να αποφασίσω. Πάντως. Κοιτάξτε, μια άλλη ιδέα. Ε, γιατί όχι ποδήλατο, γιατί για να έρθετε από την Κομισιόν ε, στο Κοινοβούλιο δεν θα μπορούσατε κάλλιστα να χρησιμοποιήσετε ποδήλατο. Θα μπορούσα μάλιστα να ποδηλατήσω μαζί σας. Εγώ στην Κοπενχάγη ζω 9 χιλιόμετρα μακριά από το γραφείο μου και συχνά χρησιμοποιήσω το ποδήλατο. Το ξέρουν οι Δανείοι. Όχι μόνο γιατί είναι φιλοπεριβαλλοντικό, αλλά και γιατί είναι καλό τρόπο για να ξεκαθαρίσει λίγο έτσι το μυαλό σου. Και το πρωί και το βράδυ. Βέβαια βλέπω ότι ενώ στην Κοπενχάγη, ας πούμε, εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα να κάνω ποδήλατο και να έρθω ε, από το σπίτι μου στο γραφείο και να κάνω αυτή τη διαδρομή με ποδήλατο αυτά τα 9 χιλιόμετρα. Εδώ στο, στις Βρυξέλλες δεν υπάρχουν τόσοι πολλοί ποδηλατόδρομοι και τα λοιπά τόσα πολλά ποδήλατα. Ε, κοιτάξτε, όχι, θα πάμε πολύ καλύτερα στο Βέλγιο με τα ποδήλατα από ό,τι νομίζει ο κόσμος. Ε, θα πρέπει να το δοκιμάστε. Η επόμενη ερώτηση. Από τα ποδήλατα πάμε στο Μεξικό, γιατί εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι χρειαζόμαστε μια νομικά μια νομικά δεσμευτική λύση στο Μεξικό στο τέλος του χρόνου. Πρέπει να μιλήσουμε με μία ενιαία φωνή, αλλά πρέπει να ανακτήσουμε την ηγετική στάση που έχει η Ευρώπη και απογοητευόμαστε που δεν θα ζητήσετε το μείον 30. Μπορείτε να πείτε μείον 30% με κάποιο, κάποια υποσημείωση. Με αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον μπορείτε να δείξετε την ηγετική στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τονίσατε ότι ο κύριος στόχος σας είναι να συνδέσετε τα συστήματα εμπορίας εκπομπών της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά στην Κοπενχάγη ήταν σαφέ ότι αν εστιάζαμε μόνο στην αμερικάνικη θέση από την ευρωπαϊκή πλευρά στην Κοπενχάγη, οδήγησε σε αποτυχίες και όχι σε πρόοδο. Πώς λοιπόν θα αντιμετωπίσετε μια συμμαχία των θεληματικών κατά κάποιο τρόπο με χώρες όπως είναι η Βραζιλία και η Ινδία στα πλαίσια του ΟΗΕ για μια λύση η οποία θα είναι δεσμευτική για όλους. Στο τέλος αυτού του, για το τέλος αυτού του μήνα. Αυτό το οποίο είπα είναι ότι δεν θα πάρω κάποια απόφαση. Εγώ δεν είμαι υπουργό στη Δανία πια, δεν θα είμαι επίτροπο παρά μόνο ενδεχομένω αργότερα. Δεν μπορώ να πω τίποτα λοιπόν για το τέλο του μήνα. Αυτό το οποίο είπα είναι ότι το πιθανότερο είναι ότι θα είναι 20% με κάποιες προϋποθέσεις πηγαίνοντας στο 30%. Αυτό είναι ρεαλιστικό, αυτό μάλλον θα συμβεί και είναι πολύ καλύτερο από αυτούς που λένε ότι ναι να το βάλουμε στα 25% ή να μείνουμε μονάχα στο 20%. Γιατί ορισμένα κράτη-μέλη έχουν παρουσιάσει τέτοιε απόψεις για το θέμα αυτό σε πρόσφατες διαπραγματεύσεις. Ελπίζω ότι μέχρι το Μεξικό φυσικά θα είμαστε στο 30%. Αυτό είναι και ο σύνολο στόχος μας. Και πρέπει να διατηρήσουμε το στόχο να μην αυξηθεί η θερμοκρασία πάνω από δύο βαθμούς. Αν η Ευρώπη δεν πάει στο μάξιμου στα 30% και δεν το κάνουν και οι άλλοι και ενδεχομένω να έχουν πιο φιλόδοξους <clears throat> στόχους για το τι θα γίνει μετά το 2020, δεν θα παραμείνουμε κάτω από το όριο των δύο βαθμών πρόσθετη θερμοκρασία. Αυτό είπαμε ότι ήταν ο στόχος μας στην Κοπενχάγη. Έχουμε μία ευθύνη να το κάνουμε αυτό και τώρα πρέπει να εφαρμόσουμε τα συμπεράσματα αυτής της απόφασης. Αν θέλουμε να μείνουμε κάτω από τους δύο βαθμούς, θα πρέπει να εφαρμόσουμε τις απαραίτητους, τους απαραίτητους στόχους. Υπάρχουν και ορισμένοι οι οποίοι θα πούν ότι η όλη διαδικασία της ε, διαδικασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήτανε δεν ήταν αρκετά επιτυχής. Εμείς δεν μπορούμε να κατασπαταλήσουμε όλες αυτές τις προσπάθειες που έχουν κατα, ε, καταβάλει τα σχέδια εθνικής προσαρμογής, τα σχέδια ευελιξίες. Έχουμε ένα τεχνολογικό πλαίσιο του οποίου γνωρίζουμε τα στοιχεία, ξέρουμε τα στοιχεία του πλαισίου προσαρμογής. Δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε όλα αυτά. Τώρα ξεπερνάω το χρόνο, δεν μπορώ να σας πω περισσότερο, αλλά πιστεύω ότι είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην καταλήξει το συμπέρασμα ας ξεχάσουμε το σχέδιο του ΟΗΕ και το πλαίσιο του ΟΗΕ. Αυτό είναι υπερβολικά απλό συμπέρασμα και θα μας οδηγήσει σε τεράστια απώλεια χρόνου. Συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να υποστηρίξουμε πλήρως τη διαδικασία του ΟΗΕ μέσα στο 2010. Αλλά όταν έχουμε τώρα αυτές τις ε, μορφές συμφωνιών όπω η Κοπεχάγη που είναι υποσχέσει σε μεγάλο βαθμό, πώ είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρξουν διπλές καταμετρήσεις από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Μήπως θα ήταν καλύτερο να θέσουμε στόχους εσωτερική μείωση των εκπομπών για να μην υπάρξει επικάλυψη στους στόχους και διπλή καταμέτρηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε να μην κάνουμε διπλή καταμέτρηση. Και οι αναπτυσσόμενες χώρες ανησυχούν πολύ περισσότερο γι' αυτό από ότι οποιοδήποτε άλλο. Λένε ωραία με τους ε, μηχανισμούς σα αυτού οι οποίοι είναι ευέλικτοι, αλλά αν μονάχα προχωρούμε σε μείωση εκεί που είναι εύκολο μονάχα και στη συνέχεια πρέπει να επιτύχουν κάτι επιπλέον. Πώς θα συναρμοστεί αυτό με τις εθνικές τους δράσεις, αυτό θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα και θα πρέπει να προσπαθήσουν όλοι να βρουν μια καλή λύση για το θέμα αυτό, γιατί οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία <clears throat> στα θέματα αυτά. Δεν θέλουν να καταπλέψει μια στρατιά από ελεγκτές και λογιστές να μετρήσει και να τους πει τι ακριβώς κάνουν. Είναι πάρα πολύ λοιπόν τεχνικά πεπλεγμένο το θέμα αυτό και ιδίως στον τομέα της δασοκομείας. Αν κάνουμε λοιπόν μια συμφωνία στο, Μεξι... στο Μεξικό, αυτό θα πρέπει να είναι ένα από τα πράγματα τα οποία θα πρέπει να α, ληφθούν υπόψη μέσα στους στόχους του 2012 και επέκεινα. So it's fine to support the UN, uh, we would agree, but uh, Τότε συμφωνούμε για να υποστηρίξουμε τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά χρειάζεται ομοφωνία 192 ετών. Υπάρχει αναλλακτικό σχέδιο. Ακόμα και για το Μεξικό δεν υπάρχει συνένεση. Αυτό είναι το ερώτημα. Αν υπάρχει καλή συμφωνία, τότε το Σουδάν δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα την τελευταία στιγμή. Πρόεδρος, όμως είναι μη ρεαλιστική αυτή η συμφωνία, όπως και το να έχουμε 192 χώρες να συμφωνούν. Θα δούμε. Κύριος Φρέντρικ Κυρία Φρέντρικ ευχαριστώ. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, το ότι μιλάω τελευταία είναι δύσκολο γιατί όλα υπόθηκαν. Πάντως το χαρτοφυλάκιό σας είναι το καινούριο στοιχείο αυτής της Επιτροπής. Πολλά αναμένουμε από εσά και είναι πολλές οι προσδοκίες. Όπως και ο συνάδελφος μέχρι, και η συνάδελφος μέχρι τώρα με έχετε εγωιτεύσει γιατί δυόμιση ώρες τώρα είδαμε την εθελοντική σας θέση, την θέλησή σας και δεν είμαι δανή αντίθετα με τη συνάδελφο. Ήδη απαντήσατε σε πολλά ερωτήματα που είχα κατά νου και μεταξύ αυτών και το ερώτημα για αυτό τη δυσκολία της οριζόντιας αρμοδιότητας που έχετε και τελικά δεν είναι διάλογος που θα πρέπει να κάνετε με τους άλλους ε, συναδέλφους σας αλλά μάχη να δίνετε σας ρωτώ λοιπόν εγώ τι θα γίνει με τις σχέσεις σας προς τα έξω. Δεν αναφερθήκαμε καθόλου στις σχέσεις με τον Μπαράκ ε, Ομπάμα και τον Χουτζιντάου. Πώς ε, θα ε, συνεργαστείτε με τον πρόεδρο Μπαρόζο για αυτόν τον διάλογο. Δεν κατάλαβα το τελευταίο σας ερώτημα. Πώς θα συνεργαστώ. Κάτι σε διεθνές επίπεδο δεν κατάλαβα. Τα είπα και εγώ λίγο γρήγορα πώς με αυτούς τους δύο κύριους παίκτες, είπα και Κίνα, θα επιβάλλετε τις απαιτήσει σας όταν αυτό απαιτεί και συνεργασία και με τον πρόεδρο Μπαρόζο. Απάντηση. Νομίζω ότι κάτι που εγώ που μπορώ να προσφέρω σε αυτή τη θέση είναι η εμπειρία μου. Έχω φίλους και γνωστούς με τις αντιπροσωπείες όλων των χωρών. Νομίζω ότι με τον Κινέζο αντιπρόσωπο ξοδέψαμε εβδομάδες. Πολλές Κυριακές περάσαμε μαζί. Νομίζω ότι τον συνάντησα δέκα φορές μέσα στο 2009. Γνωρίζω λοιπόν τους διαφόρους ανθρώπους και θα προσπαθήσω να διαδραματίσω όσο γίνεται πιο ισχυρό ρόλο μπορώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, προετοιμαζόμενοι τώρα για το Μεξικό υπήρξαν πολλές προκλήσεις. Είχαμε ιδιαίτερο πρόβλημα με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Στην ουσία όχι. Ξέρω τι, πώς φαίνονται τα πράγματα τώρα με την ομάδα των 77 και με το Σουδάν, όμως Έχουμε στενή συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες και ίσως αυτό είναι ένας τομέας όπου η Ευρώπη ως Ευρώπη μπορεί να ε, ενισχύσει τη θέση. Δηλαδή ε, ε, σε συνεργασία με την Αφρική, με την Ένωση των Μικρών Νήσων, ακριβώς εκεί να προωθήσει τις διάφορες προτεραιότητες. Συμπληρωματικό ερώτημα. Είναι σημαντική η επικοινωνία και βλέπουμε ότι και εσείς είστε πολύ καλοί στην επικοινωνία. Το είδαμε και στην Κοπενχάγη πέρα από τα καλά λόγια που μπορεί κανένας να πει, ε, στην πραγματικότητα είναι δυσκολότερα τα πράγματα. Πώς θα εξασφαλίσετε να συμμετάσχουν και οι πολίτες σε αυτήν την προσπάθεια. Υπάρχει σήμερα αυτή η οικονομική κρίση, πώς θα εξασφαλίσετε το ότι η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών θα είναι ανάμεσα στους προτεραιότητες όλων των Ευρωπαίων πολιτών, γιατί μας χρειάζεται η συνεργασία τους. Uh, because... Εξαίρετο το ερώτημά σας. Χωρίς καμία αμφιβολία και εξαιτία του όλου θορύβου για την Κοπενχάγη και το πώς τελικά έγιναν τα πράγματα. Τελικά πολλοί κατάλαβαν ότι υπάρχουν κλιματικές αλλαγές. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα σε σύγκριση με 3, 4, 5 χρόνια. Όλοι το γνωρίζουν πλέον και νομίζω ότι πρέπει να παραμείνει στο προσκήνιο. Και ίσως και η οικονομική κρίση ξεκαθάρισε τα πράγματα για τον κόσμο, ότι κάτι δεν πάει ίσως καλά στον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε, χρησιμοποιούμε την φύση. Θα πρέπει ίσως να ξανασκεφτούμε το τι ίχνος αφήνουμε στην γη αυτή. Οπότε υπάρχει η συνειδητοποίηση, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη υποχρέωση για όλους εμάς που εργαζόμαστε στο ευρωπαϊκό σύστημα, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Να το κοινοποιήσουμε αυτό, να το πούμε φωναχτά και δυνατά στους πολίτες. Γιατί βλέπουμε και τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat και βλέπουμε ότι αυτός είναι ένα τομέας όπου πραγματικά ο κόσμος περιμένει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ενεργή, να κάνει τη διαφορά. Και εκεί όλοι από κοινού πρέπει να επικοινωνήσουμε καλύτερα με τους πολίτες. Thank you. The Επόμενη ερώτηση. Βέσλουντ. Κυρία Βέσλουντ. Εδώ είμαι. Με λίγες εξαιρέσεις, όλα όσα είπατε σήμερα είναι πιστικά και θετικά. Αλλά είναι σημαντικό η Επίτροπος ε, για το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην έχει απλώς ε, να μην είναι ικανή στα λόγια, να είναι αποτελεσματική, να περάσει την κατάλληλη νομοθεσία. Ε, ανησυχώ λιγάκι για την έλλειψη ε, πληροφοριών από μέρου σα. Δεν, δεν μα είπατε τίποτα για το τι σκοπεύετε να κάνετε όταν αναλάβετε το αξίωμά σα. Θα σα δώσω μια ευκαιρία στο τέλο τη ακρόαση, λοιπόν, να μα πείτε συγκεκριμένα τι νομοθέτημα σκοπεύετε να θέσετε στο τραπέζι αν πάρετε το, το θόκο αυτό. Ε, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ξεχωρίσω κάτι, αλλά είπα ξεκάθαρα νομίζω ότι θέλω να κάνω ένα κλιματικό και μεταφορικό πακέτο, κάτι τεράστιο, έτσι δεν είναι λίγο αυτό. Αυτό είναι έκφραση ε, του mainstreaming, της ένταξης του κλίματος, δηλαδή σε όλες τις πολιτικές. Επίσης μίλησα για την έρευνα και την προετοιμασία των δημοσιονομικών προοπτικών. Αυτά δεν είναι λόγια και ένα περιεχομένου. Είναι δύσκολη πολιτική δουλειά αυτή για να υλοποιηθεί θα υπάρξουν πολλές πρωτοβουλίες που θα απορρεύσουν από το πακέτο ενέργειας και κλίματος και το ETS, ε, η εμπορία των εκπομπών, θα είναι μία από τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, γιατί είναι ήδη εν εξελίξη. Ε, φέτος χρειάστηκε να κάνουμε μία αναθεώρηση για τα αυτοκίνητα θα πρέπει να κάνουμε μια αναθεώρηση τα αυτοκίνητα για να δούμε πού είμαστε σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν, αυτά είναι συγκεκριμένα πράγματα, προσοχή, έτσι. Αλλά δεν έχω στη διάθεσή μου έτσι, πολλά νομοθετικά εργαλεία. Ε, ένα τμήμα τη δουλειά μου θα είναι να συνεργαστούμε εμείς, να βρούμε ιδέε για το, να διαμορφώσουμε έτσι τα επόμενα βήματα. Δεν είναι εύκολο κάτι τέτοιο, είναι δύσκολο. Αλλά μερικές φορές, μερικά από τα αποτελέσματα που ελπίζω ότι θα υπάρξουν δεν θα, θα προέρθουν κατά ανάγκη από νομοθετήματα που θα προωθήσω εγώ, αλλά θα τα προωθήσουν κάποιοι συναδελφοί μου. Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας. Ήταν εύκολο. Είναι εύκολο να μιλάμε για αυτοκίνητα, ειδικά όταν κανείς προέρχεται από μια χώρα που δεν έχει αυτοκίνητο βιομηχανία. Επομένως, ε, οι μεταφορέ είναι πολύ σημαντικές, ε, οι μεταφορέ αγαθών κτλ. Τι μέτρα θα προωθήσετε ε, για να αντιμετωπίσετε τις χερσαίε μεταφορέ. Δεν έχουμε κάνει αυτά που θα έπρεπε να κάνουμε ω Ευρωπαϊκή Ένωση για τα φορτηγά. Θα υπάρξει μια πρωτοβουλία. Ίσως θα είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που θα κάνουμε. Επίση υπάρχει αυτή η νομοθεσία για τα αυτοκίνητα. Πρέπει να αναθεωρηθεί οπωσδήποτε. Ως ε, υπουργό θυμάμαι πόσο δύσκολη ήταν αυτή η συζήτηση στο Συμβούλιο. Ε, συχνά βλέπουμε ότι η βιομηχανία διαμαρτυρείται και λέει «Α, είναι δύσκολο όλα αυτά, είναι αδύνατο». Αλλά και τελικά βλέπουμε ότι όταν προχωρούμε, προχωρούμε αρκετά γρήγορα. Από, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι πιστεύαμε και μάλιστα και πιο φιλόδοξα. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να αναθεωρήσουμε, να εξετάσουμε αν προχωρήσαμε αρκετά. Ε, γιατί είναι στο τομέα αυτοκίνητο που η τεχνολογία κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία υποψήφια Επίτροπε. Ε, εγώ δεν νομίζω ότι είναι μειονέκτημα να έρχεται κανείς στο τέλος των ερωτήσεων θα ήθελα να σταθώ στο ερώτημα το οποίο ετέθη ήδη και στα γραπτά ερωτήματα το ερώτημα της ε, συμπερίληψης των αεροπορικών μεταφορών. Δυστυχώς στην ακρόαση της Επιτρόπου τη μεταφο... του... Επιτρόπου για τις μεταφορές δεν μπόρεσα να πάρω μια απόφαση. Ίσως ε, δεν μπορείτε να απαντήσετε ακριβώς σε αυτό το ερώτημα. Το θέμα που έχω εγώ να θίξω είναι περισσότερο το θέμα της συνεργασίας με το Κοινοβούλιο. Πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι εκθέσεις πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βάσει του άρθρου 255 θα καταλήγουν σε προτάσεις της Κομισιόν. Πώς θα επηρεάσετε τον κύριο Μπαρόσο σε αυτές τις περιπτώσεις για να υποστηρίξετε τις προτάσεις του Κοινοβουλίου όταν πρόκειται για ένα θέμα το οποίο προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πώς θα το υποστηρίξετε μέσα στο Σώμα των Επιτρόπων. Ευχαριστώ κύριε Λίζε. Ξέρετε ότι υπάρχει αυτή η συμφωνία πλαίσιο η οποία πρέπει να τύχει επαναδιαπραγμάτευση μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Πρόεδρου της Κομισιόν. Γι' αυτό εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να μπω σε λεπτομέρειες. Απλώς μπορώ να σας πω ποια είναι η εμπειρία μου από το Δανικό Κοινοβούλιο και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα να μπορεί κανείς να συνεργάζεται με τους κοινοβουλευτικούς, όχι μόνο όταν έχετε ένα νομοθέτημα το οποίο πρέπει να περάσει, αλλά ακόμα και πριν φτάσει κανείς αυτό το στάδιο, δηλαδή στο στάδιο της προετοιμασίας. Μέσα στα πλαίσια της κλιματικής θεμετολογίας, αν εγώ είμαι <clears throat> εγκριθός επίτροπο, θα συνεργαστώ και μαζί σας και θέλω να το κάνω αυτό πολλές φορές και με έναν τρόπο ο οποίος είναι άτυπος γιατί μπορεί κανείς να έχει μια στρογγυλή τράπεζα με διάφορους εμπλεκόμενους, κάποιοι από τους οποίους είναι βουλευτές. Αυτό μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα των θέσεων οι οποίες θα προέρθουν και θα είμαι πάντα ανοιχτή στις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχει πάντα μια γενική πολιτική, αλλά χρειάζεται και η συμμετοχή του Κοινοβουλίου και μια καλύτερη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά είμαι πάντα ανοιχτή στι επικοδομητικέ προτάσει ήδη από τα πρώιμα στάδια οποιασδήποτε πρόταση νομοθετική, την οποία θέλουμε να κάνουμε. Ευχαριστώ. Αυτό είναι μια γενική δέσμευση, αλλά θέλω να σας ρωτήσω πιο συγκεκριμένα. Υπάρχει μια ε, διαδικασία για την διαθεσμική συμφωνία που θα διαπραγματευτεί ο κύριος Μπαρόσο με το Κοινοβούλιο. Αλλά θα ήθελα απλώς να σας ενθαρρύνω να πείσετε τον κύριο Μπαρόσο να ακολουθήσει τον δρόμο τον οποίο θέλουμε εμείς και να σας ζητήσω κατά πόσο στο ρόλο σας εσείς ως υποψήφια Επίτροπος θεωρείται ότι όταν το Κοινοβούλιο ακολουθώντας μια συγκεκριμένη διαδικασία καταλήγει σε μια πρόταση, θα πρέπει να την υιοθετεί η Κομισιόν και αν δεν το πράξει θα πρέπει να έχει αποχρόντες λόγους για να μην το πράξει. Μα έτσι ακριβώς είναι. Πρέπει να έχει κάνει πολύ καλούς λόγους για να μην ακολουθήσει μια τέτοια πρόταση. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας είναι σαφές ότι υπάρχει απόλυτη ισότητα μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου σε ένα ευρύτατο χώρο θεματολογίες. Γι' αυτό πρέπει να βρούμε νέους τρόπους για να επωφεληθούμε αμοιβαία από αυτή τη νέα κατάσταση και να συνεργαστούμε περισσότερο. Νομίζω ότι το σύνολο ευρωπαϊκό εγχείρημα θα ευνοηθεί ιδιαίτερα από το να είμαστε πιο ορατοί σε θέματα που εμπλέκουν άμεσα τους πολίτες μας και γι' αυτό εσείς ως εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών πρέπει να εμπλέκεστε σε αυτές τις διαδικασίες. Αγαπητοί συνάδελφοι, φτάσαμε στο τέλος του γύρου ερωτήσεων και απαντήσεων. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας και Μεταφορών για τις ερωτήσεις τους και φυσικά την κυρία Χέντεγκάρτ για, τα, για τις απαντήσεις σας. Όπως είπε πρέπει να είναι και διασκεδαστική η προστασία του κλίματος. Και είδαμε πως στην Κοπεχάγη με τεράστιο ενδιαφέρον, με τεράστιο ενθουσιασμό πάρα πολλοί άνθρωποι είτε μέσα στον χώρο της διάσκεψης ή ακόμα και έξω παρακολουθώντας από την τηλεόραση εκατομμύρια άνθρωποι παρακολουθήσαν με μεγάλο ενδιαφέρον την διαδικασία της Κοπενχάγης και επομένως έχουμε ένα θέμα που είναι σημαντικό για πάρα πολλούς και για το κοινό. Ελπίζω, πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η συμφωνία, αυτή η συζήτηση μάλλον σήμερα ήταν πράγματι διασκεδαστική και συναρπαστική και ήταν πληρέστατη και εκτενής εγώ δεν χρειάστηκε καν να χρησιμοποιήσω το σφυράκι μου σήμερα. Αλλά μετά από την, τις προηγούμενες ακροάσεις είδα ότι δεν υπήρχε λόγος να περιορίσω την κυρία Χέντεγκαρτ, η οποία πολλές φορές μίλησε σχεδόν έξω από τα δόντια, ήταν πάρα πολύ ειλικρινής και ανοιχτή. Χρειάζεστε λοιπόν αυτή την ικανότητα πυθούς χρειάζεστε αυτήν την δέσμευση, χρειάζεστε να έχετε μια γερή ραχοκοκαλιά γιατί δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσει κανείς τέτοιες εγκάρσιες αρμοδιότητες. Εγώ είμαι σίγουρος από τη δική μου πλευρά ότι εσείς μπορείτε να το κάνετε και θα εξασφαλίσετε αυτές τις αρμοδιότητες. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Αλλά <clears throat> αυτό που είναι σημαντικό είναι να εξασφαλίσουμε ότι αυτά τα οποία δεν επετέθηκαν στην Κοπενχάγη και αυτά τα οποία θα είναι επιτάπητος στις 31 Ιανουαρίου από του, τα μέλη του ΟΗΕ, αυτά δεν φτάνουν για να περιορίσουμε την αύξηση θερμοκρασία σε δύο βαθμούς. Μας φέρνουν στους τρεις ή τέσσερις βαθμούς αύξηση θερμοκρασία. Έχουμε ενώπιον μας ένα τεράστιο εγχείρημα τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα και όχι λιγότερα. Αν λοιπόν εσείς εγκριθείτε ως επίτροπος. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα έχουμε ένα επίτροπο, μια επίτροπο η οποία θα είναι δυναμική και δεσμευμένη. Και τώρα έχετε το λόγο για τις τελικές σας παρατηρήσεις. Πέντε λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πραγματικά πολύ για τις ερωτήσεις σας, για την επικοδομητική ατμόσφαιρα. Είναι η πιο μεγάλη προφορική εξέταση που χρειάστηκε να περάσω στη ζωή μου, αλλά υπήρχε προετοιμασία και προσπάθησα να εστιάσω ε, στα, στις συγκεκριμένες αρμοδιότητες του χαρτοφυλακίου μου. Θα είμαι πολύ σύντομη, γιατί ούτως ή άλλως α, καλύψαμε πάρα πολλά θέματα σήμερα. Α, όπως εγώ θεωρώ και όπως νομίζω διαπιστώσατε, το, η κλιματική αλλαγή είναι η πρόκληση που αντιμετωπίσει η γενιά μας. Ναι, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Ακούσαμε για αυτά σήμερα το πρωί. Δεν θα είναι εύκολο να καταπολεμήσει κανείς την κλιματική αλλαγή. Ε, δεν είναι κάτι που γίνεται ανέξοδα. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα, το διοξύ του άνθρακα, οι τιμές, φόροι ε, κτλ. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι όσο πιο πολύ διστάζουμε να δράσουμε, τόσο πιο ακριβό θα γίνει και τόσο πιο σοβαρή θα γίνει η κρίση του κλίματος και θα αναγκαστούμε τελικά στο μέλλον να κάνουμε σοβαρότατε αλλαγέ στον τρόπο ζωή μας και εμείς και τα παιδιά μας. Επομένως, δεν υπάρχει εύκολη λύση. Αλλά πιστεύω ότι αν χρησιμοποιήσουμε ε, την ικανότητα που έχουμε να βρούμε καινούριε λύσεις, καινοτόμε, ε, τεχνολογικές, ε, θα τα καταφέρουμε. Πιστεύω ότι η περιοχή στον πλανήτη που ασχολείται με τον πιο πιστικό τρόπο για αυτό το θέμα και που θα ασχοληθεί τα επόμενα πέντε χρόνια, αυτή η περιοχή θα ευημερήσει ε, στρατηγικά, πολιτικά και οικονομικά. Ε, όσο πιο γρήγορα κάνουμε κάτι, τόσο καλύτερα. Ε, και όχι μόνο αυτό, αλλά θα μας ωφελήσει. Ε, εμείς είχαμε πρωτοποριακό ρόλο. Θα πρέπει να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, να τον κρατήσουμε. Πολλά μπορούμε να κερδίσουμε ε, από την ενεργειακή ανεξαρτησία και την ενεργειακή ασφάλεια, αν τα κάνουμε όλα αυτά που είπα σωστά. Ελπίζω να τα καταφέρουμε, να βρούμε λύσεις που θα λάβουν υπόψη ε, διαφορετικές παραμέτρους. Κλίμα, ενεργειακή ασφάλεια και δημιουργία θέσεων απασχόληση. Αυτό θα πρέπει να είναι το όραμά μας, γιατί αυτό είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να δράσουμε. Και επομένω, νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα πείσουμε και τον υπόλοιπο κόσμου, τις υπόλοιπες χώρες. Αυτό σημαίνει, σημαίνουν οι διεθνείς διαπραγματεύσεις. Κάναμε κάποια σημαντικά πράγματα στην Κοπενχάγη, αλλά όπως διαπιστώσαμε σήμερα το πρωί, έχουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Πάντως, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε τον ΟΗΕΣ, όχι σε αυτή τη φάση. δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Θα πρέπει να, φυσικά, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμα να πετύχουμε την διεθνή συμφωνία. Ε, θα πρέπει να μείνουμε άγρυπνοι, να αυξηθεί η συνείδηση στους πολίτες, να δώσουμε το καρό παράδειγμα, να τους δείξουμε τις ε, πετυχημένες ας πούμε, προσπάθειες που έχει γίνει. Νομίζω ότι έχουμε σημαντικό ρόλο να παίξουμε. Τα επόμενα πέντε χρόνια θα είναι κρίσιμα. Γι' αυτό θα ήθελα να συνεργαστούμε για να κάνουμε πραγματικότητα αυτές τις αλλαγές. Τις αξίζει η Ευρώπη, τις αξίζουν οι πολίτες και τις αξίζει ο κόσμος. Και τις περιμένουν εξάλλου οι πολίτες. Ε, Νομίζω λοιπόν ότι εσείς και εγώ ως Επίτροπος για το κλίμα και την κλιματική δράση μπορούμε να τα καταφέρουμε τα επόμενα χρόνια. Thank Σας ευχαριστούμε για αυτό το μήνυμα και έχει κλείσει η ακρόασή μας. Απλώς θα συναντηθούν οι συντονιστές μας στο 1G2 στις 12.30 για την αξιολόγηση.